Καλημέρα σας, καθίστε. Ελπίζω να περάσατε όλοι πολύ καλές διακοπές. Ξέρετε ότι η περίοδος που ακολουθεί είναι δύσκολη και ότι θα πρέπει να δώσουμε μάχη για κάθε σέντ, ε, για κάθε λεπτό. αλλάξαμε ορισμένα πράγματα τώρα ε, σε επίπεδο δημοσιονομικό. Εμείς κάναμε κάποιες διαφορετικές προτάσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Λοιπόν, περνάω στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του μηνός Ιουνίου. Μέχρι το τέλος συνεδρίασης, αν δεν έχετε αντιρρήσεις, θα θεωρηθούν δεκτά. Το σημείο 3 είναι οι ανακοινώσει της Προέδρου. Απλά θα ήθελα να σας μεταφέρω ότι γίνεται δικτυακή αναμετάδοση της συνεδρίασής μας. Επίσης σε επίπεδο γλωσσικό δεν έχουμε πορτογαλικά, λιθουανικά, βουλγαρικά και τσεχικά. Ούτε και σλοβενικά και ε, η γλώσσα της Μάλτας. Και παράλληλα όποιος θέλει να μιλήσει Ολλανδικά ναι μεν μπορεί αλλά δεν μπορεί να ακούει τα Ολλανδικά. Ελπίζω παράλληλα να έχετε όλοι μπροστά σας τις κάρτες ψηφοφορίες. Στην περίπτωση που υπάρξουν δυσκολίες στην ψηφοφορία θα τις χρησιμοποιήσουμε. Αν δεν έχετε την κάρτα στείλτε κάποιον να σας τη φέρει. Έχω μια κάρτα, αλλά έχει διαφορετικό όνομα. Εγώ θα ψηφίσω, λες και είμαι ο κύριος Παναγιώτοφ. Εντάξει, σας βαφτίζουμε για σήμερα Παναγιώτοβα. Πράγματι το θέμα ποια είμαι λέει η κυρία Πακ. Οι συντονιστές στο τέλος της συνεδρίασης θα συνεδριάσουν και το απόγευμα θα ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό 2011. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας όπως γίνεται κάθε χρόνο, θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για το σχέδιο του Γενικού Προϋπολογισμού, όπως κάθε χρόνο είπα. Για τον τομέα φυσικά για τον οποίο είμαστε αρμόδιοι. Εμείς έχουμε μία γνωμοδότηση σε δύο κατευθύνσεις. Καταρχάς έχουμε την λεγόμενη παραδοσιακή θα έλεγα, κλασική γνωμοδότηση. Δεν έχω ίσως προετοιμάσει όσο καλά χρειάζεται αυτά που πρέπει να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, από τη μία έχουμε τη γνωμοδότηση προετοιμάσει και από την άλλη έχουμε τις απόψεις μας για το σύνολο των τροπολογιών. Ο εισηγητής μας παρουσίασε το προσχέδιό του εδώ και αρκετό καιρό. Μας παρουσίασε επίσης και τις τροπολογίες τις οποίες τα κατέθετε. Έχουμε μία προθεσμία η οποία ήταν, είχαμε μία προθεσμία η οποία ήταν η 23η Ιουλίου. 88 τροπολογίες κατετέθησαν, επαναλαμβάνω 88 τροπολογίες. 24 από τις τροπολογίες αυτές ε, τις κατέθεσε ο εισηγητής ο ίδιος. θα δώσω στον κύριο Λόκεγκάρντ ε, τον λόγο να συμπληρώσει αυτά τα οποία μέχρι τώρα έχει πει. Λόκεγκάρντ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές για το πνεύμα συνεργασίας το οποίο επέδειξαν. Να ευχαριστήσω επίσης και τα μέλη της γραμματείας της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εγώ είμαι για πρώτη φορά εισηγητή και η βοήθεια των ανθρώπων της γραμματείας ήταν πολύτιμη. Ευχαριστώ λοιπόν όλο τον κόσμο για την ε, συνεισφορά του. Το να αποφασίσει κανείς για τα δημοσιονομικά, για τον προϋπολογισμό είναι κάτι το οποίο στην ουσία μοιάζει λίγο με το να φτιάχνει κανείς τον κατάλογο για τα ψώνια του. Εύκολο μεν, αλλά όχι και τόσο εύκολο τελικά. Εμείς στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής καθορίσαμε τις προτεραιότητες μας για την επιλογή των δημοσιονομικών γραμμών για τις πιλωτικές ε, δράσεις. Προσπαθήσαμε να δώσουμε προτεραιότητα στην εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Πρόκειται για μια θα έλεγα πρόταση την οποία κάνουμε η οποία αντικατοπτρίζει μια κάποια συνένεση και στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020 θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Σχετικά για τον αθλητισμό, έχουμε αρμοδιότητα και σύμφωνα με τη συνθήκη για να αναλάβουμε δράσεις εμείς ε, κάνουμε μία πρόταση για αύξηση των πιστώσεων, τα οποία, οι οποίες συγγνώμη, θα κατευθυνθούν προς τον αθλητισμό. Τα πράγματα πάνε σχετικά καλά. Προσπαθούμε να πιέσουμε και την Επιτροπή Προϋπολογισμών να μας υποστηρίξει. Ευτυχώς έχουμε συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται πάρα πολύ καλά στο εσωτερικό της Επιτροπής Προϋπολογισμών και θα βοηθήσουν. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ και την Προεδρία ε, της Επιτροπής μας για τη βοήθεια της. Η κυρία Πρόεδρος, ε, πράγματι έχουμε αποφασίσει να στείλουμε μια σκληρή επιστολή, όχι αγενή βέβαια, στους 27 ε, υπουργούς οικονομικών ζητώντας τους να σεβαστούν τις ανηλυμένες τους υποχρεώσεις και ιδιαίτερα σε περίπτωση κρίσης όπως η σημερινή η πολιτική κατάρτιση πρέπει να παραμένει ισχυρή. Έχουμε απαντήσεις τέσσερις μόνο από Ιρλανδία, Σλοβενία, Βέλγιο και Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Το Βέλγιο και η Ιρλανδία ευχαριστούν για την επιστολή μας και μας λέγουν ότι θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση αυτή. Από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία πήρα μια μακρά απάντηση όπου μου εξηγούν ε, ποια είναι η δράση την οποία θα αναλάβουν. Εν πάση περιπτώσει είναι λίγο περίπλοκο, είναι και στα γερμανικά. Είναι στη διάθεσή σας εφόσον το ε, επιθυμείτε αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να περάσετε σεμινάρια για να κατανοήσετε τέτοιου είδους επιστολές της γερμανικής δημόσιας διοίκησης. Άπτεται των αποφάσεων οι οποίες καλύπτουν μία επταετή περίοδο και στα πλαίσια της επταετούς αυτής περίοδου ε, προβλέπονται να γίνουν ορισμένες περικοπές και δεν προβλέπεται κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής να γίνουν περικοπές, αλλά βέβαια λέγουν ότι εκεί όπου τα χρήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, οι πιστώσεις οι οποίες δεν καταλήγουν, σε αυτή την περίπτωση καταργούνται για την επόμενη χρονιά. Ε, στον τομέα των δικό μας, στον κλάδο των δικό μας δεν τίθεται αυτό το θέμα, γιατί ό,τι υπήρχε διαθέσιμο το έχουμε απορροφήσει και καταναλώσει. Εν δεν καταλαβαίνω την επιστολή της Γερμανικής Δημόσιας Διοίκησης, Ευχαριστώ τον κύριο Λέκεγκαρντ, ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές, οι οποίοι και αυτοί προσπάθησαν και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία χωρίς καθυστερήσεις. Έχουμε αρκετές τροπολογίες μαζί τις οποίες, ομαδών τις οποίες μπορούμε να ψηφίσουμε. Ε, υπάρχει κάποιος ο οποίος διαφωνεί με, να ψηφίσουμε, με το να τις ψηφίσουμε όλες μαζί οι πέντε πρώτες σελίδες του εγγράφου για τον προϋπολογισμό να ψηφιστούν μαζί λοιπόν. Στην ουσία εδώ ζητάμε την αποκατάσταση των παλαιότερων πιστώσεων και εκφράζουμε την αντίθεσή μας με τις μειώσεις του Συμβουλίου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις με την πρόταση αυτή, συνεπώς ποιοι είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών, τις οποίες ψηφίζουμε ομαδών, κατά αποχές Δύο καταψήφισαν, αλλά μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία διαμορφώθηκε ήδη. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ομάδα τροπολογιών, οι οποίες θα ψηφιστούν μεμονωμένα. «58-17» η πρώτη. Για νέα πολιτικά προγράμματα κινητικότητα καθηγητών. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία 1 για το διαβίου κατάρτιση. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες στο εσωτερικό. Ποιες είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, η ίδια πλειοψηφία δεκτή. Συμβιβαστική 2 για τον αθλητισμό προπαρασκευαστικές δράσει υπέρ κατά Αποχέ. η ίδια πλειοψηφία δεκτή. Κάποιοι Βρετανοί και κάποιοι Πολωνοί ήταν κατά. Λοιπόν, τώρα, 58-18. Ε, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Κατά. Κανείς. Ακόμα και ο Ήτον Χάρης. Ούτε αυτός δεν είναι κατά. Εν πάση φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. 58-23. Αλλά έχει ζητήσει ο Ήβο το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω να γίνει μια διόρθωση ε, στα ισπανικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Η λέξη reclaim στα αγγλικά να πάρει τη θέση της λέξης restore, τίποτα άλλο. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας της 5823 κατά αποχές δεκτή. 58-82 υπέρ. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία υπαρίθμου 58-82. Λοιπόν, υπερ, άρχεται η ψηφοφορία. Κοιτάξτε, έχουμε ήδη ουσιαστικά ψηφίσει. Την 5823. Και εσείς θέσατε τώρα σε ψηφοφορία την 5882. Ναι, διορθώνει η κυρία Πάκ. Ναι, πράγματι ψηφίσαμε την 5823 και τώρα ψηφίζουμε την 58 82. Απλά έγινε η παρέμβαση του Ιβο Μπελέτ. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας για την 5882. Απορρίπτεται. Τώρα η επόμενη Σάντσε Σμιτ υπέρ 5884. Κατά. Παρακαλώ, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Schließe die Abstimmung. Εγκρίνεται 19 υπέρ 8 κατά και μία αποχή. Προφορική τροπολογία. 1. Τάκουλα Χάγκλουντ. Τάκουλα. είπαμε να το βάλουμε ως σχόλιο. Okay. Κατά. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 10 υπέρ 16 κατά. 58-21 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αυτή εδώ. 5 και 3, 8. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Α, θέλετε τσεκ. Ωραία. 58-88 ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται 58-54. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58-25. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5873 58 58-73 αυτή εκπίπτει η 58-53 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58-56 αυτή εκπίπτει καλώς η 58-08 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εκπίπτει η 5866, Η 58-57 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5858 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ παρακαλώ να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 58-59 Μακλάκιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58-60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58-28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58.00 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58.61 α αυτή εκπίπτει καλά η 62 τότε 58.62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58.63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58-64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58-65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58-67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Η 58-37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58-68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58-32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58-69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58-33 υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5870 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5871 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. 5872 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5874 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5875 υπέρ. Κατά. Εδώ χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τελείωσε. Εγκρίθηκε 17 υπέρ 12 κατά. «58-39 υπέρ». Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58-76. Εκπίπτει. 58-40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επομενη εκπιπτη εκπίπτει. 58-42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58-78 εκπίπτη 58-43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επομενη εκπιπτη εκπίπτει. 58-51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επομενη εκπίπτη εκπίπτει ή 58-81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58-85 υπέρ κατά... Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα για να είμαστε βέβαιοι. Αρχίζει. Εγκρίνεται λοιπόν με 15 υπέρ 13 κατά. 58-89 έχει αποσυρθεί. 58-90 κύριε Βέλετ. Αν δέχεται η ε, κυρία Ματέρα να βάλουμε μια μικρή προφορική τροπολογία, μείωση από τα 5 εκατομμύρια στα 1,8. Επομένως μια δραστική μείωση. Η πρόεδρος. Εγώ κάποια άλλα πράγματα είχα πληροφορηθεί. Ναι, είναι ακριβώς όπω το είπε ο Ήβο, διότι δεν μπορέσαμε να το μεταφέρουμε σε άλλη τροπολογία. Εγώ χθε είχα προτείνει να ενταχθεί στην τροπολογία Μπέλετ και Παλιαδέλη για τον τουρισμό κλπ. Γιατί δεν είναι δυνατόν, επειδή δεν θέλει υπήρξαν προβλήματα, διότι το συζητήσαμε και με τους άλλους συναδέλφους και με τους σοσιαλιστές και υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε όλη την προστίκη σε άλλη τροπολογία. Okay. Κώστα. Κυρία Κώστα. Νομίζω ότι στην τροπολογία που εγκρίναμε πριν, για μια νέα στρατηγική για τον πολιτιστικό τουρισμό, μια τροπολογία που παρουσίασα εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Έγινε αρκετή δουλειά και με άλλους συναδέλφους και με άλλες επιτροπές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τροπολογία αυτή, που είναι μια προσθήκη, την άκουσα χθε για πρώτη φορά. Ε, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να επισημάνουμε τη σημασία της αρχιτεκτονικής ε, ε, στα πλαίσια της προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού. Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε μια επισήμανση. Δεν θα ήθελα όμως αυτή η τροπολογία η οποία προσθέτει πολλά κονδύλια σε ένα άλλο σχέδιο το οποίο νομίζω ότι δεν γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι ακριβώς θα περιλαμβάνει είναι ένδειξη μιας κάποια σύγχυση. Δεν ξέρω λοιπόν αν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμεί σε αυτή την τροπολογία. Η πρόεδρο, κυρία Πακ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία της κυρίας Ματέρα. Ψήφι υπέρ. Με την προφορική τροπολογία που μειώνει στο 1,9. Η κατά. Απορρίπτεται.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 προτείνω προφορική τροπολογία για την 8 που λέμε για τους να βάλουμε ένα νέο κονδύλι και να λέει τονίζουμε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα γραμμή του προϋπολογισμού επειδή η υλοποίηση θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω των ε, υφιστάμενων προγραμμάτων κινητικότητας. Και εμείς θέλουμε τώρα να βγάλουμε το κινητικότητα ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για το ότι δεν θέλουμε να υπάρξει νέα γραμμή του προπολογισμού. Ζητάμε λοιπόν να διαγραφεί η λέξη κινητικότητα που κάνει τα πράγματα έτσι λίγο πιο σαφή. Ναι, διότι έχουμε περισσότερα προγράμματα από μόνο τα ε, κινητικότητα και το Comenius είναι και παραπάνω από κινητικότητα και μόνο. Το citizenship επίση είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Μην βάλουμε λοιπόν μόνο mobility programs, να πούμε προγράμματα γενικότερα που σημαίνει για την εκπαίδευση και την νεολαία κλπ. Σας ευχαριστώ για την ε, διευκρίνηση αυτή. Ποιος είναι υπέρ της 8. Κατά. Κανείς. Εγκρίνεται λοιπόν.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 αποχές εγκρίνεται. για τη 18. Μια μικρή φραστική τροποποίηση. Ζητούμε να διαγραφεί για τις σημαντικές μειώσεις που έχει κάνει η Επιτροπή να διαγράψουμε εκεί που λέει που έκανε η Επιτροπή γιατί είναι συζητήσιμο εάν μιλούμε όντως για περικοπή Κρατάμε λοιπόν την λέξη reductions, περικοπές, αλλά ζητούμε να διαγραφούν οι λέξεις που λένε ότι τις έκανε η Επιτροπή, η Κομισιόν. Ανησυχώντας... Λοιπόν Made by the Commission. He's not naming the one who is doing it. Καλά λοιπόν. Είμαστε λοιπόν ευγενεί απέναντι στην Κομισιόν γιατί χρειαζόμαστε. Ψήφι υπέρ τη ε, τροπολογία αυτή χωρί τι λέξει by the Commission. Κατά εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η τελική ψηφοφορία θα γίνει ονομαστικά, αρχίζει. «21 υπέρ, 2 κατά». Εγκρίνεται. Α, τη κυρία Βερζιά. Ε, δεν λειτουργεί το μηχάνημα, άρα επομένω 23, 23, 24 το κύριο Καβαντάς. Ας ξανακάνουμε. Για πατήστε τα κουμπιά τέλο πάντων. Αρχίζει η ψηφοφορία. Την ξανακάνουμε. Δεν μπορώ να σας πω ποιο κουμπί θα πατήσετε βέβαια. Εγώ απέχω. Κλείνω λοιπόν τώρα. 26 υπέρ 2 κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Λόκεγκάτ και στους ε, Σκιώδης. Και μην λησμονούμε και το προσωπικό. Ο Ρίτιγκερ τα έκανε ε, όλα πολύ καλά. So let's come to European heritage. Λοιπόν, η πρώτη νομοθετική θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα είναι το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχουμε λιγότερες νομοθετικές τέτοιου είδους ε, εκθέσεις σε σχέση με τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Όλα αυτά για λόγους επικουρικότητας Τίθεται λοιπόν το θέμα αυτό αρκετά σημαντικό. Ξέρετε ότι αυτή σε εισαγωγικά η ετικετοθεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης είχε ξεκινήσει επί Γαλλικής Προεδρίας σε εντελώς εθελοντική εθνική βάση. Τα πράγματα τώρα έχουν πάρει μια διαφορετική μορφή και έχουμε να κάνουμε με μια πραγματική πρωτοβουλία και όχι μια απλή διακυβερνητική δράση. Παρακαλώ λίγη ησυχία η παρακαθήμενη, εδώ κάνετε φασαρία μεγάλη. Η κυρία Παλιαδέλη λοιπόν είναι η συγγήτριά μας. Δεν γνωρίζω ακριβώς αν εν το μεταξύ έχετε λάβει κάποιες περισσότερες πληροφορίες οι οποίες να δείχνουν ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Εγώ έλαβα σαν παράδειγμα ένα βρετανικό έγγραφο όπου με πολύ σκληρά λόγια λέγουν ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι παράλογη, ότι δεν έχει κανένα νόημα. Ότι υπάρχουν ε, τέτοιου είδους ετικέτες σε εισαγωγικά της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο και τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι απαράδεκτες. Αντίστοιχες απόψεις ομολογώ ότι άκουσα και από την γαλλική γερουσία αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ε, έρχεται ε, σαν κάτι το οποίο θα μας εκπλήξει αυτή η αντίδραση και αυτές οι απόψεις οι οποίες ακούγονται και σε άλλες χώρες ίσως. Λοιπόν, ας δούμε ε, τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Είμαι αρκετά περίεργη να δω τι θα κάνει η κυρία Παλιαδέλη και ποιες είναι οι προτάσεις τις οποίες θα κάνει που ίσως να λάβουν υπόψη αυτές τις ανησυχίες των μεν και των δε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να καλημερίσω τους συναδέλφους και να ευχηθώ καλή και δημιουργική χρονιά εννοώντας έναρξη της καινούργια σεζόν. Ε, πραγματικά και εγώ έχω, και εγώ έχω ε, διαβάσει απόψεις ε, από μέρους κρατών μελών, τη Γερουσία, τη Γαλλική, για το Αγγλικό δεν ήξερα, ε, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να απαντηθεί με, το, με ένα ερώτημα – μας ενδιαφέρει η κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά ως εργαλείο για την ε, ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής ή όχι. Όσοι υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται ένα τέτοιο σήμα, ε, μάλλον δηλώνουν την άποψή τους ότι αδιαφορούν πλήρως για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την συνοχή της. Ε, έχω ήδη καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό την έκθεση και ελπίζω ότι αρκετοί από τους συναδέλφους έχουν διαβάσει και την οτιολογική έκθεση και το κείμενο δηλαδή της αιτιολογίας και τις ε, ε, ε τροπολογίες που προτείνω, μερικές από τις οποίες ε, ανάγονται στη λογική και άλλες που είναι πολύ πιο επιμέρους λεπτομεριακές. Είναι ωστόσο σαφές ότι η διαμόρφωση μιας κοινή πολιτιστικής ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην προσπάθειά τους να πετύχουν ευρεία συνοχή και ελληνική και οι πρόσφατες εκλογές έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει αυτό. Βεβαίως και υπάρχουν άλλοι ριζοσπαστικότεροι και προφανέστεροι τρόποι να ενισχυθεί η πίστη των Ευρωπαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ηγέτες της. Ωστόσο, η γνώση της ιστορίας της Υπήρου μας, η εξοικείωση με την πολυεθνική αλλά εν τέλει κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά και η βελτίωση της εκπαίδευσης της νέας γενιάς σε ό,τι αφορά τις ιδέες και τους ανθρώπους που πορτοστάτησαν στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη γεφύρωση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Στα όργανα τα ευρωπαϊκά και τους πολίτες της. Για, στη φάση του, ε, πριν ακόμα θεσμοθετηθεί το διακυβερνητικό, διακρατικό παλαιό σήμα που εμείς καλούμαστε να μετασχηματίσουμε ε, με, με βάση την πρόταση της, της Επιτροπής μια ευρεία διαβούλευση λοιπόν με την κοινή γνώμη και μια εκτίμηση επιπτώσεων είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ε, το διακυβερνητικό παλαιότερο σήμα θα μπορούσε να επιτύχει, καλύτερα τους στόχους του αν λειτουργούσε ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περισσότερο σαφή κριτήρια και αποτελεσματικότερο σύστημα παρακολούθησης. Ε, καταρχήν να δηλώσω ότι ασπάζουμε απόλυτα την πρόταση της Επιτροπής να αξιοποιήσει το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς ως ένα από τα μέσα για να φέρει πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Ε, κατά συνέπεια η απόφαση των καρτών μελών ε, εκτιμώ ε, και να μετατρέψουν το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς και να το εντάξουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πιστεύω ότι θα συμβάλλει στην αύξηση της προβολής του σήματος, του κύρους του σήματος, αλλά και της αξιοπιστίας του, εξυπηρετώντας και πάλι τον κεντρικό στόχο που είναι η συνοχή και η ελληνική. Αρχικά πίστευα ότι, ε, ε, ή μάλλον οραματιζόμουν θα έλεγα με αυτή την αφορμή, ένα σήμα που θα μπορούσε να υπερβεί τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να περιλάβει εντός του τουλάχιστον τη γεωγραφική έννοια της Ευρώπης και να χρησιμοποιηθεί επομένως ως ένα φιλόδοξο μέσο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε στόχους της κοινή εξωτερικής μας πολιτικής. Ωστόσο, σε μια δεύτερη ανάγνωση και έχοντας συζητήσει αρκετά με εκπροσώπους και της Επιτροπής και του Συμβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειών διαπίστωσα ότι δεν ήταν σε αυτή τη φάση ρεαλιστικό ένα τέτοιο σήμα που θα απευθυνόταν στην Ευρώπη ως Ήπειρο και όχι στην Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση θα ήταν αποτελεσματικότερο το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς να περιοριστεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υποστηρίξει καταρχήν τον στόχο του, την πολιτική συνοχή των κρατών μελών και την εμβάθυνση της κοινωνικής και πολιτιστικής σύγκλησης των λαών της. Σε ένα δεύτερο επίπεδο αυτό το σήμα θα μπορούσε να διευρυνθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου στις οποίες, οι οποίες αναγνωρισμένα συνέβαλαν και στην ιστορία και στον πολιτισμό της Υπήρου, της Ευρώπης και γιατί όχι, ακούστηκε και αυτό σε μια από τις συζητήσεις, θα μπορούσε και να αξιοποιηθεί ακόμη περαιτέρω να διευρυνθεί και σε περιοχές εκτός Ευρώπης ως Υπήρου προκειμένου να τιμηθούν μνημεία, ιδέες, τόποι κλπ που εφάρμοσαν, αξιοποίησαν ή ε, σεβάστηκαν ε, αξίες που γεννήθηκαν στην υπηρό μας. Αλλά στην παρούσα εισήγηση αντιμετωπίζουμε το νέο σήμα ε, στην πρώτη του μορφή. Δηλαδή το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, για τις χώρες που, την, που ανήκουν σε αυτήν. Στην παρούσα εισήγηση λοιπόν θεωρούμε το σήμα όχι ως μετασχηματισμό του παλαιού αλλά ως ευκαιρία για την αξιοποίηση της εμπειρίας του παλαιού προκειμένου να το ξαναδούμε συνολικότερα. Για το λόγο αυτό, πρώτον, προτείνουμε την μετονομασία του σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου ο τίτλος αυτός να ανταποκρίνεται στον πρωταρχικό στόχο όπως τον ε, είπα λίγο πριν, ως μέσο δηλαδή για τη συνοχή και την αλληλεγγύη πρωτίστως ή τουλάχιστον σε πρώτη φάση ανάμεσα στους πολίτες των κρατών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, θεωρήσαμε αναγκαίο να, να, να προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου λογότυπου που θα διαφοροποιεί το νέο σήμα από το παλαιότερο του διακρατικού χαρακτήρα. Ε, για το λόγο αυτό, ως πρόταση, ε, από, σε συνέχεια μάλλον αυτής της λογικής, τρίτον προτείνουμε να καταργηθούν οι σύνθετες μεταβατικές διατάξεις που περιγράφονται στο άρθρο 18 της πρότασης, επειδή θεωρούμε ότι τα δύο σήματα θα μπορούν να συνεπάρξουν δυνητικά στον ίδιο τόπο, επειδή ο, ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν στηρίχθηκε σε διαφορετικά εν τέλει κριτήρια. Δηλαδή ένα ένα κράτος, ένας τόπος, συγγνώμη, ένα μνημείο να έχει και το παλαιό σήμα που έλαβε στη φάση που το σήμα ήταν διακρατικό αλλά βεβαίως να, μπορεί να λάβει εφόσον καλύπτει τα κριτήρια του νέου σήματος και το καινούριο σήμα. Τα δύο σήματα να συνεπάρχουν. Τέταρτον, προκειμένου να διαφυλάξουμε το κύρος του σήματος από μια σχεδόν γραφειοκρατική λογική ισοκατανομής πόσες χώρες, πότε θα γίνουν, πόσα, πόσοι αριθμοί θα προκύψουν με τόπους που διεκδικούν και θα λάβουν εν τέλει το σήμα και για να δώσουμε περισσότερο χρόνο και στην προεπιλογή και στην τελική επιλογή δηλαδή σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και κυρίως για να διασφαλίσουμε ένα σοβαρό σύστημα παρακολούθησης να δούμε δηλαδή αν τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέχθηκαν οι τόποι ε, εξακολουθούν να εφαρμόζουμε προτείνουμε όχι την διαδικασία αναέτος αλλά ανά δύο χρόνια αυτό θα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μπορούμε να τα αλλάξουμε αργότερα, θα, ανακούφι, θα μας έδινε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σοβαρότερα την πρώτη φάση εφαρμογής του. Ε, πέμπτον, σε ό,τι αφορά τους διακρατικούς χώρους, δηλαδή χώρους που επιλέγουν δύο κράτη να, α, ε, ε, να προτείνουν ως υποψήφια για την απονομή αυτού του τίτλου, ε, συμφωνούμε με την πρόταση της Επιτροπής να ευνοούνται, δηλαδή να προηγούνται θα λέγαμε στην επιλογή, και ως προς την ποσόστοση ακριβώς επειδή υποστηρίζουν τη λογική των κοινών στοιχείων, τη δημιουργία δικτύων και βεβαίως ενισχύουν και ενθαρρύνουν τη συνεργασία ανάμεσα σε κράτη ή σε περιφέρειες. Μόνο για πρακτικούς λόγους θεωρούμε ότι ένα κράτος μέλος από τα δύο που θα, ή τα τρία που θα ε, συνυποβάλλουν μια τέτοια πρόταση ως υποψήφια να λάβει το σήμα θα πρέπει να λειτουργεί ως συντονιστής στις συζητήσεις και με την ομάδα εμπειρογνωμόνων και την Επιτροπή. Ομολογώ ότι αναζήτησα τρόπους να ενισχύσω το ρόλο της ομάδας των εμπειρογνωμόνων αυτών που θα κάνουν την τελική επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα προτείνουν μάλλον την τελική επιλογή ε, σε ό,τι αφορά στην απονομή ή την ανάκληση του σήματος. Νομικά όμως κάτι τέτοιο το ψάξαμε δεν είναι δυνατό αλλά παρόλα αυτά στην εισήγησή μας προτείνουμε μια ουσιαστικότερη συνεργασία της ομάδας αυτής των εμπειρογνωμόνων με την Επιτροπή, με ενημέρωση, συστάσεις, διαβουλεύσεις κλπ. Περισσότερο ακόμη μας απασχόλησε, <clears throat> ομολογώ, ε, μας απασχόλησαν τρόποι για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία και της απονομής και της ανάκλησης. Νομικά όμως κάτι τέτοιο φαίνεται ότι είναι δυσχερές ε, επειδή δεν είναι δυνατόν να έχει περισσότερες αρμοδιότητες από εκείνους που, περιγράφονται, καταγράφονται στην ε, πρόταση της Επιτροπής. Όμως εναλλακτικέ δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την καλύτερη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήταν να γνωμοδοτεί για την επιλογή των χώρων, αυτό θα επιβράδυνε πολύ δραματικά την διαδικασία. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει πλήρη κατάλογο των προεπιλεγμένων χώρων και να ενημερώνει το Συμβούλιο και το, Ευρωπαϊκό, το, και Κοινοβούλιο. Αυτό θα παρήχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωβουλευτές, επαρκή χρόνο να αντιδράσουν σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια προβλήματα που προκύπτουν. Όγδον, Θεωρήσαμε απαραίτητη τη συμμετοχή στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων ε, ενός μέλους της Επιτροπής Περιφερειών ε, ώστε να δώσουμε φωνή σε ένα θεσμό που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και που ασχολείται και με τον πολιτισμό. Ένατον, κάναμε σαφέστερα τα κριτήρια με επιμέρους διατυπώσεις που περιλαμβάνουν τους νέους, τον τουρισμό. <coughs> Could you Thank you. Τα άτομα με αναπηρίες κλπ. Και, και θεωρήσαμε αναγκαίο να αποσαφηνίσουμε όρους. Αυτό είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Όπως ιστορία και πολιτισμός της Ευρώπης, και οικοδόμηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφοροποίησαμε δηλαδή τον όρο Ευρώπη από τον όρο Ευρωπαϊκή Ένωση στο κείμενο το συγκεκριμένου. Τέλο, προτείνουμε τη δυνατότητα οικειοθελού αποχώρηση, α πούμε, επιστροφή του σήματο, προκειμένου χώροι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην εφαρμογή των κριτηρίων να μπορούν με δική του πρωτοβουλία να αποσύρουν το, το, το, το ε, σήμα. Όχι μόνο να του το πάρουν, επειδή δεν τα εφαρμόζουν, αλλά και ήδη να δηλώσουν την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές. Ολοκληρώνοντας την προφορική αυτή <clears throat> εισήγηση, θεωρώ υποχρέωσή μου να δηλώσω ότι το σήμα από μόνο του δεν μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί ωστόσο να συμβάλλει μαζί με άλλες πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση του, του συγκεκριμένου ζητήματος. Δηλώνω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά χωρίς τη συνεργασία της Γραμματείας της Επιτροπής Πολιτισμού και τις επαφές μας με τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου και βεβαίως χωρίς τους πολύτιμους επιστημονικούς συνεργάτες μου. Προσβλέπω στις παρατηρήσεις και τις απόψεις σας, περιμένω με αγωνία ομολογώ τις τροπολογίες σας και ελπίζω πως με τη στενή συνεργασία μας τις επόμενες εβδομάδες θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο μέγιστη δυνατής αποδοχής για ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είπε και ε, η πρόεδρος ε, της Επιτροπής μας που θα αντανακλά τις κοινέ ε, θέσεις μας πάνω στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία συνάδελφε. Ιδιαίτερα εκτεταμένη η πρώτη αυτή, η παρουσίασή σας μάλλον σίγουρα θα υπάρχουν ερωτήσεις από μέρος των συναδέλφων. Κύριε Μπόρις. Ευχαριστώ για μια πραγματικά αναλυτική και λεπτομερέστατη παρουσίαση. Είναι λοιπόν σαφές ότι η εμπειρία της UNESCO είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και από ό,τι φαίνεται αναπτύσσονται ορισμένες μορφές τουρισμού ε, στην Ευρώπη ιδιαίτερα όπου οι περιηγητές αναζητούν συγκεκριμένους χώρους τους οποίους έχει σηματοδοτήσει η UNESCO στα πλαίσια ορισμένων θα έλεγα παραδοσιακών πολιτιστικών δικτύων και υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι πολύ ενδιαφέροντες χώροι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται πάντα στα κριτήρια της UNESCO αλλά είναι σημαντικοί για την ιστορία της Ευρώπης. Συνεπώς λοιπόν η προσπάθεια της εισηγητρίας είναι πολύ θετική γιατί μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε το σήμα αυτό και για συνοριακές περιοχές. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιοχές ενδιαφέροντος ανάμεσα στις χώρες μας και αυτό επιπλέον δείχνει θα έλεγα τη δυνατότητα και για κάποια μαθήματα ιστορίας, γιατί από τη μία τα σύνορα μετακινούνται, από την άλλη οι συγκεκριμένοι χώροι παραμένουν πάντα μάρτυρες ενός συγκεκριμένου παρελθόντος. Λοιπόν, μπορούμε να βοηθήσουμε την κατανόηση της ιστορίας της Ευρώπης μέσα από την χορήγηση τέτοιου είδους σημάτων. Υπάρχει μια περιοχή στην Ευρώπη, ένα μικρό παράδειγμα να θέσω τώρα, είναι τα καθολικά τάγματα. Τα καθολικά τάγματα έχουν δημιουργήσει ε, στους, ε, στην Ευρώπη εξαιρετικά ε, μοναστήρια, εξαιρετικές μονές σε όλη την Ευρώπη. Και να σαν παράδειγμα ένα τέτοιο δίκτυο πολιτιστικών επισκέψεων το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει, στην, να δημιουργήσει ένα δίκτυο, θα έλεγα, επισκέψεων και να προκαλέσει πανευρωπαϊκού τύπου ενδιαφέρον. Ε, εάν συνδυάσω αυτά που περιλαμβάνετε εσείς στην εκθεσή σας και τα όσα είπε τώρα λίγο ο κύριος Μπόρης, και αν τα συνδυάσω με τα όσα ψηφίσαμε σήμερα το πρωί, όπου τονίσαμε ιδιαίτερα ότι μας ενδιαφέρουν οι πολιτιστικές οδοί και να ανοίξουν και νέε, που είναι στην πραγματικότητα θεσμοί, αν θέλετε, που τους εμφύσισε πνοή ζωή το Συμβούλιο της Ευρώπης, που όμως έχουν μεγάλη σημασία. Και εμείς θέλουμε να υπάρξουν ακόμη περισσότερες. Και το γεγονός ότι θα υπάρχουν οι δυνατότητες τώρα να γίνονται αιτήσει για τη χορήγηση του σήματος και για υπερμεθόριες περιοχές ή διαμεθοριακές, διαμεθοριακών ενδιαφέροντος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μπορούμε έτσι να ξυπνήσουμε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας για τις οδούς αυτές. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά διασυνδέονται τα πράγματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για τα όσα έκανε και όλες τις ε, ανησυχίες που προσπάθησε να λάβει υπόψη, κυρίως για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον προπολογισμό και να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εργασιών που έχουν ήδη γίνει. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο περισσότερα ή δυνατόν ως προς τα κριτήρια επιλογής και ποιος ε, θα είναι υπεύθυνο για την επιλογή. Διότι αν θέλουμε να έχουμε ε, μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, παρά το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία επιλογής, δεν θα πρέπει από την άλλη να είναι στοιχείο ανταγωνισμού ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους που να φέρουν το σήμα, διότι ε, έτσι θα χαθεί ο κοινό στόχος μιας κοινή ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Πώς μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και κοινό ενδιαφέρον να συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη και όχι να ανταγωνίζονται μεταξύ των. Προσφάτως, το ιστορικό κέντρο του Άμστερνταμ πήρε το σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και πολλοί από τους πολίτες δυσαρεστήθηκαν. Και αυτό γιατί ε, όταν ένας χώρος ε, λαμβάνει το σήμα της UNESCO, υπάρχουν περιορισμοί για τις ε, αρχιτεκτονικές βελτιώσεις, τα νέα κτίρια ή τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κέντρο μιας πόλης. Εάν ε, λοιπόν ε, μιλάμε για το κέντρο μιας ευρωπαϊκής πόλης, έχουμε πάρα πολλές ε, δραστηριότητες εκεί, δεν έχουμε μόνο επισκέψεις τουριστών, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι δημόσιοι χώροι και θα ήθελα να ξέρω λίγο περισσότερα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζεται αυτό. Ποιες θα είναι οι συνέπειες πέρα από το σήμα αναγνώριση ω πολιτιστική κληρονομιά θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στη χρήση των ε, χώρων αυτών ώστε να διατηρηθούν. Ναι, μεν είναι λογικό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια ισορροπία, ιδίω όταν ε, υποτίθεται ότι ε, θα πρέπει να συνδέονται με την ευρωπαϊκή ιστορία και την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά μέσω αυτού του σήματο. Και έχω και μια τελευταία ερώτηση Υπάρχει τρόπος ε, να συνδέσουμε άλλα προγράμματα όπως το Ευρωπαϊάννα, το οποίο θέλει να έχει ένα ψηφιακό κατάλογο των ευρωπαϊκών πολιτιστικών ε, στοιχείων και πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε αυτά ώστε να εκπαιδεύσουμε και τους νεότερους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και τον, ε, το σύνολο του πληθυσμού για τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά προϊόντα. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Επισημαίνω όμως ότι δεν υπάρχει, υπάρχει μάλλον πύλη για τα πολιτιστικά και εκεί βάζει και η Κομισιόν ό,τι επιθυμεί. Φύσας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν η ιδέα μου φαίνεται πάρα πολύ καλή. Ε, στην πείρα που είχα ως ε, Υπουργός Αυτόνομης Περιοχής ε, ήμουν αρμόδης για πολιτιστικά θέματα και καταλαβαίνω πόσο σημαντικός είναι ο πολιτιστικός τουρισμός. Και αυτό φυσικά ευνοεί και την ε, μόρφωση και την εκπαίδευση όλων των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά φυσικά βοηθά και την οικονομία. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν αρκεί να υπάρχει ένα σήμα σε ένα μνημείο. Καταρχάς θα πρέπει το μνημείο αυτό, ε, ο χώρος αυτός να βρίσκεται σε, καλές, σε καλή κατάσταση. Ποιος θα το ελέγχει αυτό. Αυτή τη στιγμή σε ένα μνημείο είναι κληρονομιά της UNESCO. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εποπτεύουν, επιτηρούν ώστε ο χώρος αυτός να είναι σε καλή κατάσταση και ορισμένες φορές υπάρχει δυνατότητα απόσυρσης του σήματος εάν δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και ορισμένες φορές διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν μνημεία που βρίσκονται σε πολύ καλή κακή κατάσταση. Ποιος λοιπόν θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο, ε, διότι μπορεί να υπάρχει ένα μνημείο το οποίο θα έχει το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και μπορεί να βρίσκεται σε πάρα πολύ κακές ε, συνθήκες και καταλαβαίνετε ε, ότι εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν ένας έλεγχος και θα πρέπει να υπάρχει και κάποια προϋπόθεση ώστε να είναι αυτά τα μνημεία αποδεκτά σε όλη την Ευρώπη γιατί αλλιώς δεν θα χρησιμεύει σε τίποτα το σήμα. Επίσης να πω ότι εμένα δεν μου φαίνεται λογικό η κάθε χώρα να έχει τον ίδιο αριθμό μνημείων ή να μπορεί να προτείνει τον ίδιο αριθμό μνημείων. Με όλο το σεβασμό το Λουξεμβούργο δεν είναι το ίδιο με τη Γερμανία ή την Ισπανία ή την Ελλάδα ως ε, κατηγορία, ως ε, αριθμό μνημείων που περιλαμβάνουν και επομένως όπως γίνεται και με την UNESCO θα πρέπει το σήμα αυτό να γίνεται με βάση τη σημασία των ίδιων των μνημείων και όχι επειδή θα πρέπει να έχουν ίσο αριθμό μνημείων όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Η Μαρή Τερέζη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Que nous avions euh, élaboré Euh, je pense faudrait que nous nous penchions sur sa proposition de ίσως πρέπει πράγματι να σκεφτούμε αυτό το οποίο είπε η συγγήτρια να, εξ, να αλλάξουμε τον τίτλο, την, το όνομα του σήματος αυτού. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι αντιπροσωπεύει. Προτείνει με ένα σήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Παλιαδέλη. Είναι μια καλή ιδέα, αλλά από την άλλη ίσως ε, να διαφοροποιείται λίγο το σήμα αυτό από το σήμα έτσι όπως το φανταζόμασταν που θα κάλυπτε το σύνολο του πολιτισμού της Ευρώπης. Θα ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων πριν πάρουμε κάποια απόφαση. Τώρα, σχετικά με την συχνότητα απόδοσης του σήματος αυτού, η κυρία Παλιαδέλη λέει ότι θα πρέπει να δίδεται σε διετή, αναδιετία ε, και αυτό πρέπει να το δούμε πάλι. Τώρα για τις μεθοριακές περιοχές έχει σημασία το να ζητάμε να γίνεται η επιλογή από τις χώρες μεμονωμένα θα επιβαρύνει τη διαδικασία. Αν θέλουμε να πετύχει το σήμα αυτό, θα πρέπει οι διαδικασίες να είναι οι απλούστερες δυνατές, οι προσβασιμότερες πιο εύκολα σε όλους τους ενδιαφερομένους και γι' αυτό τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ε, γνωστά. Εδώ η πληροφόρηση και η ενημέρωση θα παίξουν τεράστιο ρόλο. Κυρία Μπαντία ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ από την πρώτη μέρα που παρουσίασε η Επίτροπος αυτή την πρωτοβουλία, κατάλαβα ότι δεν αναφερόμαστε απλώς και μόνο σε μνημεία έχουμε κατά νου συνέχεια όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό σήμα πολιτιστικού τουρισμού, σκεφτόμαστε μνημεία, πέτρες, κάστρα, εκκλησίες. Νομίζω ότι εγώ αντιλήφθηκα ότι αυτό πήγαινε λίγο παραπέρα και από τη συζήτηση που ακούω σήμερα μου φαίνεται ότι όλοι επικεντρωνόμαστε για άλλη μια φορά σε πέτρες. Εγώ κατάλαβα ότι μιλούσαμε για χώρους, θα μπορούσε να είναι ένα δάσος, θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε, που έχει κάποια σημασία ε, ως προς την οικοδόμηση της Ευρώπης που δημιουργεί αναμνήσεις, μνήμες και ούτω καθεξής. Ήθελα απλώς να το διευκρινίσω διότι μου δόθηκε η αίσθηση ότι επικεντρωνόμαστε μόνο στον πολιτιστικό τουρισμό, επίσκεψη μοναστηριών, κάστρων, εκκλησιών, μουσείων. Θα έπρεπε να έχουμε λίγο πιο ανοιχτού ορίζοντες και να βλέπουμε λίγο παραπέρα από αυτά. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ. Um, Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω την τροπολογία 6 για το άρθρο 2. Διαβάστε την αν θέλετε. Λέει για τους σκοπούς της αποφάσεως αυτής μνημεία στο, επίσης χώροι σε αστικό ή υπεθρό, σε αστικό τοπίο ή υπεθρό και περιλαμβάνει επίσης πάρα πολλά άλλα ακόμα και άειλο πολιτιστικό αγαθό το οποίο συνδέεται με ένα συγκεκριμένο χώρο θεωρούνται και αναφέρονται ως χώροι. Νομίζω ότι ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που ζητείς. Άρα περιλαμβάνεται ήδη μέσα. Η κυρία Παλιαδέλη ήδη έχει συμπληρώσει με τα ε, αυτά, με αυτά την επιφάνεια των υδάτων δηλαδή. Θέλουμε δηλαδή βασικά αυτό που θα προστατεύεται να μπορεί να το δει κανεί. Όμω υπάρχουν και αυτά που δεν φαίνονται, δεν είναι ορατά, ωστόσο είναι υπαρκτά και θα πρέπει και αυτά να μπορούν να λαμβάνουν ε, το σήμα αυτό. Ε, και βέβαια αυτοί που θα απαρτίζουν την Επιτροπή θα καθίσουν να σπάσουν τα κεφάλια τους, να βρουν τρόπο ώστε να μπορεί να απονεμηθεί το ε, σήμα αυτό. Η κυρία Πάντς της Επιτροπής. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται θετικά απέναντι στην έκθεση αυτή και ευχαριστεί την κυρία Παλιαδέλη για μια εξαιρετική προσπάθεια. Οι αλλαγές που προτείνονται έχουν σαν στόχο να κάνουν πληρέστερο αλλά και πιο ευκρινές το κείμενο η έκθεση λοιπόν είναι συμβατή με τις γενικές ανησυχίες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε η πρωτοβουλία αυτή να έρχεται συμπληρωματικά άλλων πρωτοβουλειών και να μην επικαλύπτεται με αυτές. Και επίσης θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι το πρόγραμμα αυτό ελαφρύ σε επίπεδο διαχειριστικό εννοούμε και να είναι επίσης ε, όσο περισσότερο ορατό από το ευρύ κοινό γίνεται. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτή η πρώτη πρόταση αποτελεί μια πάρα πολύ καλή λύση για να πετύχουμε όλα αυτά. Να διευκρινίσω ίσως κάποια θέματα τα οποία ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κάτι το οποίο ίσως να βοηθήσει. Για την επιλογή των συγκεκριμένων θέσεων τοποθεσιών να σας παρασέμψω στο άρθρο 7. Το άρθρο 7 πράγματι διευκρινίζει τα κριτήρια. Η επιλογή θα πρέπει να γίνεται σε δύο φάσεις και αυτό διευκρινίζεται στο έγγραφο. Θα υπάρχει μία προεπιλογή σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη θα είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κριτήριο και το δεύτερο θα γίνεται μέσω η δεύτερη επιλογή μέσω ενός ευρωπαϊκού πάνελ σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο θα ελέγχει μάλιστα αν τα κριτήρια εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο στο σύνολο της Ευρώπης. Βέβαια θα μπορούν οι εθνικές αρχές να κάνουν μια διπλή πρόταση σε μια περίπτωση και εκεί το Ευρωπαϊκό Πάνελ θα επιλέγει τη μία από τις δύο. Τώρα σχετικά με την UNESCO και η αναφορά που έγινε στο κέντρο του Άμστερνταμ και της χρήσης του δημοσίου χώρου στις πόλεις. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρότασή της δεν περιλαμβάνει τέτοιου είδους λεπτομέρειες και κανόνες. Το πνεύμα αυτό της, της, αυτού του σήματος παραμένει διαφορετικό από την UNESCO. Μιλάμε για το συμβολισμό που μπορεί να έχουν τοποθεσίες και ε, μέρη σε σχέση με την ιστορία της Ευρώπης. Δεν μιλάμε για διατήρηση, για συντήρηση, για τεχνικά θέματα που αφορούν τον, τουρισμό και, τον τουρισμό και γι' αυτό και δεν επιβάλλουμε κανένα περιορισμό. Είναι θέμα εκπαιδευτικό περισσότερο. Υπάρχει επίσης και ένα άλλο θέμα, οι τοποθεσίες αυτές θα πρέπει να συντηρούνται σωστά και εδώ η αρχή της επικουρικότητας φυσικά ισχύει. Πέραν αυτής όμως υπάρχει πάντα και στο άρθρο 7 για τα κριτήρια, το τρίτο τμήμα του άρθρου 7 περιλαμβάνει την ανάγκη να υπάρχει σωστή διαχείριση των συγκεκριμένων προεπιλεγμένων χώρων και προβλέπεται μια διαδικασία παρακολούθησης, θα έλεγα ελέγχου, που θα διεξάγεται και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πάνελ, έτσι ώστε οι τοποθεσίες αυτές να συντηρούνται σωστά. Σε σχέση με τις δραστηριότητες οι οποίες θα διεξάγονται εκεί κτλ. Και σαν τελική θα έλεγα λύση μπορεί να υπάρχει και αφαίρεση σήματος, αλλά είναι μια μακρά διαδικασία. Λοιπόν, ε, νομίζω να κάλυψα κάποιες από τις απορίες ουσίας. Να πω ότι είμαστε απόλυτα διαθέσιμοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την εισηγήτρια και προς τους κοιόδης εισηγητές εφόσον επιθυμούν. Και θα συνεχίσουμε, ελπίζω, από κοινού την προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει. Η Πρόεδρος Πακ, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο σχόλια, αν με επιτρέπετε. Εάν προβλέπετε να γίνονται προτάσεις των χωρών μελών. Θα έχουμε μετά μια κριτική επιτροπή που θα επιλέγει. Το ερώτημα είναι εάν προταθεί ένας μόνο χώρος με την ευρύτατη έννοια. Χώρος με την ευρύτατη έννοια. Θα είναι δύσκολο να γίνει επιλογή. Θα έπρεπε λοιπόν να θεωρηθεί ως όρος εκ των ονού κάνευ να γίνονται τουλάχιστον δύο προτάσεις από κάθε χώρα ώστε να μπορεί να γίνεται και κάποια επιλογή. Εάν προτείνεται ένας χώρος και με αυτόν δεν συμφωνεί καθόλου η Κριτική Επιτροπή, θα πρέπει να μπορεί να τον απορρίπτει. Άρα θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε οι χώρες μέλη να καταβάλουν προσπάθεια να επιλέγουν χώρους που να είναι πραγματικά άξιοι να λάβουν το σήμα αυτό. Και όχι να φτάνουν να απορρίπτονται από την Κριτική Επιτροπή διότι δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες. Και όπως και με την πολιτιστική πρωτεύουσα θεωρώ και εγώ ότι πρέπει και στην περίπτωση αυτή να προτείνονται τουλάχιστον δύο υποψηφιότητε. Τώρα υπάρχει και ένα άρθρο που λέει ότι μπορούν και μετά χώροι να αποφασίσουν ότι παρετούνται του σήματος. Δηλαδή μπορεί να το λάβουν σήμερα το σήμα, αλλά σε πέντε χρόνια μπορούν να αποφασίσουν ότι δεν το θέλουν. Θα πρέπει τότε να το ανακοινώσουν στην Κομισιόν και η Κομισιόν, όπω προτείνει η κυρία Παλιαδέλη, θα πρέπει να το ανακοινώσει στην Κριτική Επιτροπή. Υπάρχει όμω και ένα άλλο άρθρο εδώ που λέει καθαρά και πώ μπορεί να αφαιρεθεί το σήμα. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνε δηλαδή ώστε και να μπορεί να αφαιρείται το σήμα, η σφραγίδα και εδώ κάπως απαντούμε και στην κυρία Σάκε, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι το σήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς θα είναι τόσο αυστηρό, θα έχει τόσο αυστηρές προϋποθέσεις όπου το σήμα της UNESCO. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε τόσο πολύ αυστηροί, διότι ενδέχεται να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά από καλό. για περίπτωση όπου, για παράδειγμα, χτίζεται κάτι μέσα σε ένα χώρο όπου δεν θα έπρεπε γιατί είναι προστατευόμενος από το σήμα αυτό, ε, τότε θα πρέπει να δείχνεται κάποια ανοχή. Δεν είμαι, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ ικανοποιημένη με την αλλαγή του ονόματος. Νομίζω αυτό πρέπει να το επανεξετάσουμε, εάν δηλαδή θα γράψουμε μόνο Ευρωπαϊκό σήμα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή μόνο, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το περάσουμε ως μήνυμα. Πάντως είμαι ανοιχτή. Αν υπάρχουν άλλες προτάσεις, πολύ ευχαρίστω να τις συζητήσουμε. Παρακαλώ, εσείς κύριε Παλιαδέλη έχετε πάλι το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλούμε, μικρόφωνο. Απαντήθηκαν από, τις, ε, από την εκπρόσωπο του, ε, της, της Επιτροπής ε, να ευχαριστήσω την ε, κυρία Ικούτσετ για την ε, επιστροφή στην ουσία αυτού του σήματος ότι στην, δεν πρόκειται για ένα υποκατάστατο της UNESCO άλλα, άλλα είναι τα σήματα που, δίνει, που απονέμει η UNESCO και άλλα είναι αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνουν συμβολικά χαρακτηριστικά μπορεί να εκφράζουν να, να σχετίζονται με μνημεία που εκφράζουν ιδέες και όχι, παραδείγματο χάρη, τα ανθρακοριχεία. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα αντικείμενο μια τέτοια ε, απονομής ή μετατροπή τους σε κάτι άλλο. Ή, ε, για να θυμίσω πόσο σημαντικό είναι ότι η κατάργηση της θανατικής ποινή σημαίνει για πρώτη φορά στην Πορτογαλία. Βάζω δύο ακραία πράγματα, αλλά η ιδέα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο δεν συμπίπτει ούτε απολύτω με το cultural με τις πολιτιστικές διαδρομές, ούτε από αυτή την άποψη. Συμπληρώνει ενδεχομένως το ένα το άλλο. Ε, δεν, δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι σίγουρο. Η, το, ο χώρος πρέπει να είναι έτοιμος ή να ετοιμαστεί προκειμένου να καλύψει τα κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 7 και στα οποία θα ήμουν ευτυχής αν είχατε επιπλέον παρατηρήσεις να κάνετε με τις τροπολογίες σας. Ε, υπάρχει ένα ζήτημα με την παρατήρηση που έκανε η κυρία Πάξη ό,τι αφορά ότι είναι απαραίτητο να έχουμε δύο τουλάχιστον υποψηφιότητες από κάθε κράτος προκειμένου καθένα από τα, από τα 27 να, να πάρει το δικό του. Ε, εγώ θα ήμουν ευτυχής στο δηλώνω και ξέρετε καλά από ποια χώρα προέρχομαι <laughs> ε, θεωρώ ότι κανονικά θα μπορούσαν μερικά κράτη να μην πάρουν παρόλο που έχουν ε, καταθέσει υποψηφιότητα γιατί οι χώροι τους οποίους πρότειναν δεν καλύπτουν τα κριτήρια του σήματος. Μπορούν να βελτιωθούν και να το κάνουν αργότερα. Αυτό θα ήταν αν θέλετε λιγότερο γραφειοκρατικό, περισσότερο ουσιαστικό. Αλλά μπαίνει και μια διάσταση πολιτική που δεν θα ήθελα εγώ προσωπικά να την αγγίξω. Ε, ωστόσο, εκτιμώ, διαβάζοντας πριν ακόμη έρθω στην Ευρωβουλή, ή μάλλον με αφορμή την έλευσή μου στην Ευρωβουλή και διαπίστωσα ότι ο όρος Ευρώπη είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο μας μπερδεύει. Ο στόχος για την αλλαγή του τίτλου ε, ανταποκρίνεται, αν θέλετε κυρία Πρόεδρε, μόνο στο πρώτο κομμάτι αυτής της εφαρμογής. Έχω πολύ φιλο... θα, ήμουν, ε, θα ήταν πάρα πολύ φιλόδοξο όχι να χρησιμοποιήσουμε τον όρο Ευρώπη για κάτι που δεν είναι όλο δικό μας, ένα κομμάτι είναι και εκτός Ευρώπης, έτσι δεν είναι αυτή τη στιγμή, εκτός γεωγραφική Ευρώ, Ευρώπης, αλλά να μπορούμε να βγούμε και έξω από αυτήν. Να μπορούμε δηλαδή να απονείμουμε αυτό το σήμα και στην, σε χώρε τη νότια Αμερικής, παραδείγματο χάρη, που έχουν κάνει πράγματα ή σε ιδέε που έχουν εφαρμοστεί ε, με βάση τι ευρωπαϊκέ αξίε, όπω γεννήθηκαν εδώ. Ε, αν το θέμα είναι πολιτικό εκεί το συζητούμε αλλά εκτιμώ ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να απονέμουμε ως Ευρώπη ένα σήμα που απονέμεται στην ουσία που έχει συλληφθεί ε, ως ιδέα και απονέμεται από μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί έχω, έχω μια μεγάλη έτσι, δυσκολία να το ε, αποδεχτώ αλλά θα το δούμε. Ε, περιμένουμε με μεγάλη αγωνία τις ε, τροπολογίες σας. Δεν ξέρω μήπως δεν απάντησα σε κάποιες από τις ε, παρατηρήσεις σας. Παρακαλώ όμως να διαβάσετε την έκθεση. Ε, αξίζει τον κόπο που σας έρθουν και άλλες ιδέες που συμβάλλουν στην βελτίωση αυτής της πρότασης που έχει κάνει η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι 23 Σεπτεμβρίου, 12η μεσημβρινή, έχουμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε τροπολογίες. Επαναλαμβάνω 23 Ενάτου το μεσημέρι. Στις 27 Οκτωβρίου επιθυμούμε να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Παλιαδέλη. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερησίας διατάξεως που είναι οι πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εισήγηση είχε αναλάβει η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τον ηγετικό σας ρόλο στο θέμα αυτό. Ανυπομονώ να μάθω ποιοι συνάδελφοι θα συμμετέχουν στην σύνταξη αυτής της έκθεσης. Είμαστε στην αρχή και νομίζω ότι μας πιέζει ο χρόνος, διότι ε, μετά από τη θέση ισχύ της ενδείξης της Αβώνας, αλλά και μέσω των νέων οδηγών, οδηγιών της UNESCO και των εκθέσεων που έχουμε, είναι κατεπήγον να σκεφτούμε τις ε, πολιτιστικές διαστάσεις ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει να βλέπουμε δηλαδή την Ευρώπη ως παγκόσμιο παίκτη και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία και αν δούμε τα πολιτιστικά προγράμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι γνωρίζουμε εδώ στην αίθουσα ότι δεν θέλουμε απλώς να έχουμε έναν και μόνο πολιτισμό, αλλά αυτή την ποικιλομορφία θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε και να την αναπτύξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Roughly, I believe we could look at, at culture. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα προγράμματα αυτά με δύο τρόπους. Έχουμε καταρχάς τις εγγενείς αξίες που συνδέονται με τον πολιτισμό, στη δημιουργικότητα, στις τέχνες, ε, διάφορα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών που ε, έχει ε, ξεκινήσει η Ευρώπη αντιλαμβανόμενη αυτό το ρόλο και επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως μέσω της πραγωγής ε, των ευρωπαϊκών αξιών, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, αλλά και προσπαθώντας να συμφιλιώσουμε και να λάβουμε υπόψη τις πτυχές της ασφάλειας. Οι πολιτιστικές πτυχές φυσικά είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη θέσεων εργασίας και θέλουμε φυσικά να υπάρχει καινοτομία ως σημαντική πτυχή της παιδείας. Αφενός λοιπόν έχουμε ένα πυλώνα που πρέπει να τον ε, ε, συνδράμουμε και ταυτόχρονα υπάρχουν οριζόντια και πάρα πολλές άλλες δράσεις. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να συνδυάσουμε σε αυτή την έκθεση και να δούμε από συνολική σκοπιάς. Έχοντας λοιπόν κατά νου τη συνθήκη της Λισαβόνα, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε τέτοια προγράμματα και πώς μπορούμε να τα αναπτύξουμε με το βέλτιστο και πιο αποτελεσματικό τρόπο, ε, να υπάρχει πρόσβαση στα πολιτιστικά προϊόντα, παγκόσμια πρόσβαση η οποία θα είναι ανοιχτή στους πολίτες, να υπάρχει προϋπολογισμός ο οποίος ε, θα λειτουργεί αποτελεσματικά χωρίς πολλή γραφειοκρατία και επίσης να εξετάζουμε και τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στον τομέα του πολιτισμού. Θα εξετάσουμε λοιπόν λίγο το συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των υφιστάμενων προγραμμάτων, τα πολυστηριστικά προγράμματα, τα πολλά προγράμματα που έχουμε ανταλλαγών, το Erasmus Mundus, το Ευρωπαϊκά, τη συνθήκη της UNESCO, αλλά και θέματα πολυγλωσσίας και επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε και θέματα στα οποία ο πολιτισμός ε, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, όπως για παράδειγμα τα πνευματικά δικαιώματα, τα προγράμματα γειτονίας, καθώς και στοιχεία ε, δημόσιας διπλωματίας. Θα ήθελα λοιπόν να συνεργαστούμε και να αναλύσουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε, πώς μπορούμε να τα συντονίσουμε, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνοχή, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και ποια στοιχεία δεν θα καλύπτονται ε, ώστε να συμμετάσχουν και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο, στην κοινωνία των πολιτών, ε, ώστε η Ευρώπη να διαδραματίσει έναν υπεύθυνο και ελκυστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες διαστάσεις και τις διεθνείς σχέσεις ε, από πολιτιστικής σκοπιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Φλικενστάιν. Πρόεδρε, μετά από αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Σάκε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αν θέλετε τη δημιουργία, μια σημαντική προσπάθεια μάλλον, στην οποία η πολιτιστική πολιτική οφείλει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις και ο πολιτισμός πρέπει από μόνος του να πάρει τη μορφή ε, ενός βελτιωμένου διαλόγου με άλλες χώρες και να προωθήσει γενικότερα τις επαφές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες με τις οποίες μας συνδέουν διεθνείς σχέσεις. Αυτά ακούγονται θεωρητικά όμως. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε παράλληλα ποιος είναι ο τίτλος της δράσης την οποία ξεκινάμε. Στην ουσία λέμε για τον ρόλο του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης στις εξωτερικές σχέσεις και τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων. Αυτός είναι ο, συγκεκριμένος τίτλος. Εγώ θα ήθελα να επανέλθουμε λίγο στον αρχικό τίτλο. Βρίσκω περιοριστικό ε, τον σημερινό τίτλο αν θέλετε. Φυσικά δεν είναι προαπαιτούμενη μια μεγάλη συζήτηση επί της ουσίας και επί της θεωρίας, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε με συγκεκριμένους τρόπους ε, ποια θα είναι η συμμετοχή της πολιτιστικής, ε, αν θέλετε, πολιτικής ή του πολιτισμού στις εξωτερικές δράσεις. Ποιες είναι οι πολυπολιτιστικές ενέργειες, ποιες είναι οι πολυμερείς δράσεις τις οποίες έχουμε ήδη αναλάβει ή θα πρέπει να ξεκινήσουμε στο μέλλον και που εντάσσονται σε μια γενικότερη στρατηγική. Ποιες υπάρχουσες δομές επιτρέπουν μια τέτοια συμμετοχή του πολιτισμού στις εξωτερικές δράσεις, ποιες δομές πρέπει να δημιουργηθούν στο μέλλον έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής του πολιτισμού στις εξωτερικές δράσεις. Και τέλος, ποια είναι τα οικονομικά ή καλύτερα τα δημοσιονομικά προαπαιτούμενα για να υπάρξουν τέτοιου είδους προσπάθειες. Κυρία Παλιαδέλη ε, να δηλώσω για μια ακόμη φορά ότι θεωρώ πως ο πολιτισμός και μερικές χώρες της Ευρώπης ως χώρες και όχι ως μέλη αναγκαστικά εδώ και αιώνες έχουν, τον έχουν χρησιμοποιήσει ως ε, εργαλείο για την εξωτερική του πολιτική. Πάρα πολύ πετυχημένο. Και το βλέπουμε ακόμη και σήμερα με την Coca-Cola και τη δίσδυσή τη στην Ανατολή, τη Δύση κλπ. Είναι σίγουρο ότι ο πολιτισμός μας είναι, ε, ε ο πολιτισμός είναι εργαλείο εξωτερικής όχι μόνο δράσης και εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει επομένως να πείσουμε την Επιτροπή ότι πραγματικά πρέπει να στηρίξει ε, αυτή την ε, ε, μεριά, αυτή την όψη ενώ μιας τέτοιας πρότασης προκειμένου να αξιοποιήσει τον πολιτισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα ήθελα να γυρίσω λιγάκι πίσω προς την ε, ε, προηγούμενη συζήτηση ότι αυτό ίσως δικαιολογεί κυρία Πρόεδρε γιατί πρέπει το όρος του προηγούμενου, το σήμα του προηγούμενου ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς να αλλαγεί σε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο aggressiveness, επιθετικότητας ενεργητικής προς τα έξω, εκτός Ευρώπης, η οποία θα βοηθούσε ενδεχομένω και την εξωτερική πολιτική. Η κυρία Άστον θα έπρεπε πάρα πολύ καλά να σκεφτεί πώς θα αξιοποιήσει τον πολιτισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Βάτιμο. Ε, είμαι πεπισμένος ότι το θέμα τίθεται Υπάρχουν βέβαια νομίζω λίγο περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία ακούστηκαν μέχρι τώρα. Σαν παράδειγμα, στον κόσμο, με ποια γλώσσα θα μιλάει η Ευρώπη. Η κληρονομιά της Ευρώπης συνδέεται με τις εθνικές παραδόσεις. Οι εθνικές παραδόσεις έχουν δημιουργήσει θεσμούς, ξέρετε, πολιτιστικά Ινστιτούτα, Υπάρχουν το Γκέτε, ένα παράδειγμα δίνω, ή το Ιταλικό Ινστιτούτο σε πάρα πολλέ χώρες του κόσμου. Λοιπόν, ο πολιτισμός εισαγωγικά εξάγεται από τις, από τις χώρες, από τα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολο λίγο να το, ε, να το ευρωπαϊκοποιήσουμε σε, σε εισαγωγικά. Το θέμα της γλώσσας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα Ινστιτούτα Πολιτισμού, το Γκέτε και τα λοιπά συνδέονται κυρίως με τα μαθήματα της γλώσσας της κάθε χώρας. Οπότε με ποια γλώσσα θα βγούμε προς τα έξω σαν Ευρώπη. Με ποιο τρόπο θα δείγμαστε ομοιογενείς πολιτιστικά. Λοιπόν, η πιθανή δημιουργία κάποιων ευρωπαϊκών ε, πρωτοβουλειών για την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού στο εξωτερικό θα πρέπει να ξεκινήσει από την προώθηση και τον συντονισμό των υπαρχουσών πρωτοβουλειών των κρατών μελών. Είναι αλήθεια ότι θα υπάρξει εδώ ένα κάποιο πλεονέκτημα για κάποιες μικρές χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν τέτοια πολιτιστικά Ινστιτούτα. Αλλά ξέρετε ότι όπως και στην περίπτωση της διπλωματικής δράσης, ναι μεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρεσβείες σε εισαγωγικά στο εξωτερικό, αλλά πάντα παραμένει ο πρέσβης της κάθε χώρας αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη χώρα. Λοιπόν, υπάρχει εδώ μια δυσκολία. Πώς θα μπορέσουμε να συμπεριφερθούμε σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ξεκινήσει να εξελίσσονται και σε σχέση με τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα πρέπει να φανταστούμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Σάκε γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω το σύνολο της παρέμβασής της. Εγώ ανησυχώ από ένα κυρίως θέμα. Ο πολιτισμός για μένα είναι ουσιαστικά το μέσο ε, της ε, πολιτιστικής ποικιλότητα, ένα μέσο το οποίο βοηθάει τη συμβίωση την κοινωνική των ανθρώπων. Λοιπόν, ναι μεν θα πρέπει εμείς ε, να δείξουμε το τι είναι η Ευρώπη προς τα έξω, αλλά θα πρέπει και στο εσωτερικό της Ευρώπης αυτή την ποικιλότητα, τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, να τον δείξουμε και αυτόν έτσι ώστε να ενισχυθεί και στο ίδιο το εσωτερικό της Ευρώπης. Σαν παράδειγμα, ο σεβασμός των μειωνοτικών πολιτισμών πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ξέρουμε ότι όλοι ανησυχούμε σε αυτή τη φάση από την επιμονή κάποιων φαινομένων ξενοφοβίας. Λοιπόν, ε, η συμβίωση διαφορετικών πολιτισμών σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα μέσο πολύ αποτελεσματικό για την προώθηση του πολιτισμού. Ιδιαίτερα και στον τομέα της μετανάστευσης. Εδώ μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ μας, αλλά αν πράγματι θέλουμε να υπάρξει μια τακτή σε εισαγωγικά μετανάστευση ελεγχόμενη η οποία να λειτουργήσει ενσωματωτικά για τους πληθυσμούς αυτούς, εκεί η, ε, η αγαστή σχέση ανάμεσα στους πολιτισμούς είναι μια εγγύηση για να το πετύχει. Ο κύριος Βάτιμο ζήτησε εκ νέου το λόγο. Είναι αλήθεια ότι ένας τρόπος για να λυθούν κάποια από τα προβλήματα τα οποία έθεσα προηγουμένως θα ήταν ίσως να συνοδεύουμε, να πλαισιώσουμε την ευρωπαϊκή δράση μέσα από όργανα τα οποία να παρουσιάζουν ε, στον κόσμο ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν ας πούμε προγράμματα μελέτης ευρωπαϊκού επίπεδου και όχι μόνο εθνικού επίπεδου θα μπορούσαν να περνούν μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές. Υπάρχουν λοιπόν από τη μία οι εθνικές πρωτοβουλίες, εκεί δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές, αλλά ταυτόχρονα ας ξεκινήσουμε κάποιες υπηρεσίες ας πούμε, ε, σαν παράδειγμα προωθώντας ένα ευρωπαϊκό φεστιβάλ κινηματογράφου ή μια οι εθνικες πρωτοβουλιες εκει δεν θελουμε να κανουμε καποιες σημαντικες αλλαγες αλλα ταυτοχρονα ξεκινησουμε συνάντηση της ευρωπαϊκής νεότητας ή τέτοιου είδους ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αμυγός και όχι εθνικές. Μπορείς. Ευχαριστώ καταρχάς που άλλαξε ο τίτλος, αναφέρομαι στην εισηγήτρια εδώ. Ε, νομίζω ότι πράγματι με τον τίτλο αυτό τοποθετούμε θα καλύτερα στην εξωτερική δράση. Εγώ δεν φοβάμαι την εξωτερική δράση. Θέλω η εξωτερική αυτή δράση να είναι παρούσα χωρίς αυτό να κινδυνεύει να μειώσει την ουσία της προσπάθειάς μας. Νομίζω ότι η δύναμή μας στο εξωτερικό της Ευρώπης μπορεί να είναι ο πολιτισμός. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που έρχονται στην Ευρώπη για να δουν την Ευρώπη για το πολιτιστικό της δυναμικό, για την πολιτιστική της κληρονομιά και μόνο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να το αγνοήσουμε. Μία παρατήρηση να κάνω σχετικά με την προώθηση του ευρωπαϊκού λεγόμενου πολιτισμού στον υπόλοιπο κόσμο. Παραδοσιακά έχουμε σαν παράδειγμα τις πρεσβείες, τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών που έχουν ε, και πολιτιστικές αρμοδιότητες, οικονομικές αρμοδιότητες μεταξύ άλλων. Οι πρεσβείες αυτές πάρα πολύ συχνά ε, θα κληθούν να αντικατασταθούν στο μέλλον από την υπηρεσία κοινή εξωτερικής δράσης σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό. Οπότε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Αυτού του είδους οι ευρωπαϊκές εισαγωγικά υπηρεσίες, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του πολιτισμού. Το κόστος σε αυτή την περίπτωση θα είναι πάρα πολύ υψηλό γιατί ναι μεν σε επίπεδο διπλωματικής δράσης θα αναλυθούν πάρα πολλές ε, πρωτοβουλίες, αλλά ε, όχι πολιτιστικά, δεν προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να το συζητήσουμε αυτό. Και στα πλαίσια της συζήτησης αυτής θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και ποια είναι η πολιτιστική διάσταση αυτών των νέων υπηρεσιών που θα ασχοληθούν με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης στο μέλλον. Χάνιμπαλ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτό το θέμα. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουμε πριν προχωρήσει. Ε, καταρχήν είναι πολύ καλή ιδέα, δεν είμαι κατά, αλλά θα ήθελα να επιστήσω λίγο την προσοχή όλων σε κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να σκεφτούμε. Το πιο προφανές είναι πώς ε, προάγουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Όπως είπαν όλοι και, έχουν δίκιο, ε, το κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του πολιτισμό, ο οποίος λειτουργεί πολύ καλά με τον τρόπο που τα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ευρωπαϊκά και λειτουργούν καλά, αλλά πώς θα μεταλαμπαδεύσουμε όλα αυτά στους υπολείπους. Εγώ ακόμα δεν έχω βρει την απάντηση. Και πριν το προχωρήσουμε πάρα πολύ το θέμα αυτό, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε τι είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Διότι εγώ προσωπικώς δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα κάνουμε είναι πολύ, καλό, πολύ εύκολο να γίνει αυτό σε επίπεδο κράτους μέλους γιατί είναι σαφές τι ακριβώς θα προάγει ο καθένας. Αλλά δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό για την Ευρώπη. Η γλώσσα είναι το προφανές πρόσκομα. Όλοι είμαστε εδώ, ο καθένας ε, μας, άλλος χρησιμοποιεί ακουστικά όταν μιλάει κάποιος άλλος. Ε, η αγγλική γλώσσα είναι ίσως το πιο κοντινό που έχουμε σε μια διεθνή γλώσσα και εγώ φυσικά δεν θα ήθελα τα πάντα στο εξωτερικό για την Ευρώπη να προωθούνται στην αγγλική γλώσσα, διότι νομίζω ότι αυτό δεν είναι το πνεύμα της όλης διαδικασίας. Επίσης υπάρχει διαφορά μεταξύ εμπορική εξαγωγή ε, πολιτισμού, ε, κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ καλή η Αμερικανή. Η κυρία Παλιαδέλη αναφέρθηκε στην Coca-Cola. Υπάρχει και μουσική άλλωστε. Τα πάντα εξάγονται με πολύ εμπορικό τρόπο και μάλλον αυτό δεν είναι απαραίτητο πολιτισμός. Νομίζω ένα από τα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να εξετάσουμε είναι αντί να προσπαθήσουμε να προάγουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ως έννοια που δεν γνωρίζουμε ούτε καν και εμείς τι ακριβώς σημαίνει, να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον τοπικό πολιτισμό περισσότερο. Και ένας από τους ρόλους της υπηρεσίας εξωτερικής δράσεως θα μπορούσε να είναι να δει στις χώρες στις οποίες εντοπίζεται τι συμβαίνει εκεί και πώς μπορεί να προωθήσει τις τοπικές δραστηριότητες.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 E, chciałbym odnieść się do dwóch δύο θέμα. Ε, για τον τίτλο τώρα της ε, έκθεσης είναι το ένα θέμα και το δεύτερο θέμα είναι η, η ποικιλότητα, η πολιτισμική, η, πολυπολιτιστική διάσταση. Είναι αλήθεια η συζήτηση για τον τίτλο της έκθεσης έχει μια κάποια σημασία. Οι λέξεις έχουν ένα συγκεκριμένο όνομα και ο τίτλος μπορεί να λειτουργήσει στρατηγικά. Εγώ είμαι ακαδημαϊκός και κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής μου καριέρας μέχρι τώρα ε, πήρα μέρος στην υποστήριξη πολλών διδακτορικών διπλωμάτων και ξέρω τι σημασία έχει ο τίτλος. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του τίτλου σοβαρά γιατί θα χαρακτηρίσει τη συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό στο μέλλον. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ο Μπόρις ή ο Φλέκενστάιν. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε τώρα για την ποικιλότητα την πολιτισμική. Εδώ πρέπει να δούμε τι πρέπει να προωθήσουμε, τι πρέπει να δείξουμε προς τα έξω. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε η ποικιλία και η διαφορά μέσα στην ενότητα. Νομίζω ότι αυτά είναι λίγο θεωρητικά και πολλές φορές μιλάμε πάρα πολύ για την Ένωση και λιγότερο για την ποικιλία και για τη διαφορά. Είμαστε η Ένωση 27 κρατών, όχι 27 περιοχών, όχι 27 μειονοτήτων κρατών, ανεξάρτητων κρατών. Συνεπώς λοιπόν οι δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα ίδια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προωθηθεί ο εθνικός πολιτισμός. Δεν υπάρχει ουσιαστικά ευρωπαϊκός πολιτισμός. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί πολιτισμοί. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός κινηματογράφος, ένας ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Υπάρχει ο γερμανικός, ο πολωνικός και ο τσεχικός κινηματογράφος. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να φανούν ξεκάθαρα στη συζήτηση η οποία θα γίνει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ιδέα για την έκθεση αυτή ήταν δική μου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να την υπερασπιστώ. Πρώτων διακοπών είχα προσκαλέσει σε μια στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους οργανισμών που ασχολούνται με το με τα πολιτιστικά, όπως το Ινστιτούτο Γκέτε, το Ινστιτούτο Θερβάντες και άλλα. Και όπως δεν γνωρίζετε ορισμένοι, ήδη συνεργάζονται αυτοί σε μια ε, οργάνωση, διεθνή οργάνωση εθνικών ε, που συνδυάζει, δηλαδή που, στην οποία συμμετέχουν ε, διάφοροι εθνικοί οργανισμοί. Κανένας δεν μιλεί για μια ομοιογενή, για ένα ομοιογενή πολιτισμό. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μας συναποτελείται από την ποικιλία των επιμέρους πολιτισμών. Δεν υπάρχει λοιπόν ομοιογένεια. Είναι όμως ένας πλούτος που θα μπορούσε να είναι και μεγάλο hit, για την, ε, εξαγωγικό hit δηλαδή, για την παρουσία μας προς τα έξω, προς τον κόσμο. Και επειδή ως ευρωβουλευτές δεν ενδιαφερόμαστε μονάχα ή δεν θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε μονάχα για όλους εκείνους οι οποίοι εμφανίζουν, ε, δηλαδή για να εμφανίζουμε την Ευρώπη μονάχα ως εμπόριο, ως οικονομικά, αλλά και είμαστε και εκπρόσωποι του πιο σημαντικού μας αγαθού, δηλαδή του πολιτισμού μας. Γι' αυτό σκέφτηκα εγώ ότι κάπως πρέπει να καθίσουμε να τα μελετήσουμε λίγο αυτά. Ποια μορφή θα λάβει τώρα, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή θέλουμε να καταστήσουμε ορατή αυτή την ποικιλία των πολλαπλών πολιτιστικών εκφάνσεων. Αυτό ήταν που με ενδιέφερε. Και υπάρχουν πολλοί οργανισμοί, πολλά, πολλοί θεσμοί οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Δεν θέλουμε να εξαφανίσουμε κανένα οργανισμό ο οποίος ας πούμε εργάζεται για πολιτιστικά στη Λατινική Αμερική. Όχι. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους και να δείξουμε πώς εμφανίζεται η Ευρώπη παντού, είτε με τη φραγίδα τη Πολωνία ή με τη φραγίδα τη Γερμανία ή άλλων χωρών. Αυτά μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα. Αυτό είναι όντω ε, κάπω δύσκολο να, ε, γίνει ορατό. Είναι και λίγο δύσκολο και για μένα να το εξηγήσω. Αλλά νομίζω η δική μας υπόθεση είναι ε, να ζητήσουμε από την κυρία Άστον να τα περιλάβει τα πράγματα αυτά η οποία οι οποίοι μάλλον ασχολούνται εκεί με το ποιος, ποια εθνικότητα θα πάει πού, ποια θα αναλάβει την τάδε ευρωπαϊκή θέση και ποια την δίνα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα δεν είναι ποιος θα πάει, ποιος θα αναλάβει τη σχετική, ε, ποιος θα καταλάβει μάλλον τη σχετική θέση, αλλά να φέρει μαζί του την απαραίτητη πολιτιστική παιδεία. Και αν μπορούμε να πούμε ως Επιτροπή Πολιτισμού στην κυρία Άστον, εφόσον εσύ επιλέξεις κάποιον, μην λησμονείς ότι υπάρχουν και αυτές οι αρχές οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επιλογή. Και αν τώρα ο κύριος ή η κυρία πρέσβης δεν θέλει απαραίτητα να αναμειχθεί στον τομέα αυτό, είμαι βεβαία ότι θα υπάρχουν άλλοι, πολλά άλλα πρόσωπα που θα διοριστούν στις πρεσβείες αυτές που μπορούν να αναλάβουν το καθήκον αυτό. Άρα ας τοποθετηθεί κάποιος ο οποίος να ασχολείται με τον πολιτισμό και ο οποίος μπορεί να εμφανίσει και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μέσα σε όλη του την ποικιλία και στις χώρες αυτές όπου θα πάει. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κινηματογράφος, είναι γερμανικός, είναι ε, πολωνικός ή εσθονικός κλπ. Γιατί άλλωστε κάνουμε το φεστιβάλ αυτό με το βραβείο για τον κινηματογράφο. Ακριβώς για να τονώσουμε τον ε, ε, κινηματογράφο. Δεν θέλουμε μια, ο, ένα ομοιογενή κιανό πολιτισμό με χρυσά αστεράκια όπως είναι η σημαία. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να φανούν ανάγλυφα οι αξίες μας. Και ο πολιτισμός που έχει αναπτυχθεί μέσα από όλη αυτή την ιστορία έχει όλες αυτές τις εκφάνσεις για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι όλοι. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι το γεγονός ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί και εγγύηση, εγγύηση για την συνέχιση της ύπαρξης πολλών μικρών πολιτισμών. Το 97 μας είχε προσκαλέσει ένας Σουηδός συνάδελφος την Επιτροπή Πολιτισμού στην ε, Σουηδία, στην Κιρούνα όπου είναι το κέντρο του πληθυσμού Σάμι. Πήγαμε εκεί, τι πολύ ωραία, τι ωραία είπαμε, αλλά γιατί πάμε. Μάθαμε λοιπόν ότι εκεί ο πληθυσμός Σάμι είχε εκφράσει την επιθυμία να μας δει, για να μας ευχαριστήσει, να ευχαριστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το γεγονός ότι μπορεί και κατοικεί σε ευρωπαϊκή χώρα, σε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως με τον τρόπο αυτό προωθείται καλύτερα η πολιτιστική του ταυτότητα. Διότι με την περιφερειακή ανάπτυξη που προωθούμε υποχρώνεται και το Σουηδικό κράτος να συγχρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε και εμείς. Και έτσι με τον τρόπο αυτό ο πληθυσμό αυτός, η ομάδα, η πληθυσμιακή η ομάδα Σάμι απέκτησε πολλές ευκαιρίες να προωθήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις που την ενδιέφεραν. Εγώ λοιπόν είχα εκπλαγεί τότε πάρα πολύ ευχάριστα, διότι φάνηκε καθαρά ότι δεν, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή η οποία έρχεται να καλύψει με ένα ε, κιανό μανδύα όλο, όλα τα πολιτιστικά πράγματα, αλλά ότι δίνει την ευκαιρία να ανθίσουν και μικροί επιμέρους πολιτισμοί. Αυτή είναι στην πραγματικότητα, αυτό είναι και το μήνυμα. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε θα θέλαμε να περάσουμε και στις χώρες αυτές και ελπίζω έτσι να διασυνδεθούν και οι δικοί τους πολιτισμοί με τον δικό μας. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι το καθήκον κάποιου εμπνευσμένου ανθρώπου και αυτόν τον εμπνευσμένο άνθρωπο θα πρέπει να τον ψάξει και να τον βρει η κυρία Άστον. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Σχάκε. thank you. Um, you are a great ambassador. Ευχαριστώ πράγματι. Μπορείτε να λειτουργήσετε σαν πρέσβης του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν θα σχολιάσω. Συμφωνώ με αυτά που είπατε και με τους περισσότερους από τους συναδέλφους. Αυτή η διαφορετικότητα προφανώς και θα πρέπει να διατηρηθεί εμείς δεν μπορούμε να σκοτώσουμε ακριβώς τα βασικά θετικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, η διατήρηση της διαφορετικότητας είναι κάτι το οποίο καθιστά την Ευρώπη ενδιαφέρουσα. Υπήρξαν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις νωρίτερα. Το έφεσε ο κ. Φρέκενστάιν να δούμε τους τρόπους με τους οποίους ο πολιτισμός παίζει ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις, μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια της πρόθεσης του διαλόγου δύο χωρών ή της αποτροπής κάποιων συγκρούσεων. Πράγματι εδώ ε, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, υπάρχει επίσης γενικότερα το θέμα της προώθησης της δημιουργικότητας, και της προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών όσο γενικές και να ακούγονται όπως η δημοκρατία και η ελευθερία έκφρασης. Υπάρχουν και άλλα θέματα που τέθηκαν και ένα από αυτά αφορά τον τίτλο της πρωτοβουλίας αυτής, της έκθεσης αυτής. Έχω την εντύπωση, αλλά δεν είμαι σίγουρη, ότι ίσως να έχει δημιουργηθεί μια κάποια σύγχυση στις διαφορετικές μεταφράσεις. Στόχος της έκθεσης είναι να εξετάσουμε τις πολιτιστικές πλευρές της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει και τα νέα μέσα. Δεν θα ήθελα να αποκλείσω τα νέα μέσα γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. νομίζω ότι οι ανησυχίες που εκφράστηκαν για την εγκατάλειψη της διαφορετικότητας και της πολιτιστικής ποικιλία, αυτά νομίζω ότι έχουν καλυφθεί. Στα Ολλανδικά που κοιτάω εγώ εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής του τίτλου, αλλά δεν ελέγχω τους άλλους τίτλους στις άλλες χώρες, στις άλλες γλώσσες. Αυτά θα πρέπει να τα δείτε εσείς. Πάντως ο στόχος είναι οι πολιτιστικές διαστάσεις της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι άλλα σχόλια έχω σημειώσει εδώ. Κάποια παραδείγματα τα οποία έγιναν σαν παράδειγμα η Coca-Cola δεν είναι απόλυτα πολιτιστικό προϊόν βέβαια Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Νομίζω ότι είναι καλό παράδειγμα αυτό το οποίο δώσατε και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές σε άλλα μέρη του κόσμου, ακόμα και στο εσωτερικό της Ευρώπης και αυτή είναι η βασική θα έλεγα αρχή της συνεργασίας που θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε και πιθανές επικαλύψεις με άλλες προσπάθειες και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ελέγχουμε τις δραστηριότητες οι οποίες θα ξεκινάνε, πώς θα κυκλοφορούν οι ενημερώσεις για τις δραστηριότητες αυτές στον υπόλοιπο κόσμο, αποφεύγοντας επαναλαμβάνω με αρνητικό τρόπο τις επικαλύψεις. Το θέμα της γλώσσας. Προφανώς η διατήρηση της διαφορετικότητας και της ποικιλία περνάει και μέσα από τον σεβασμό των γλωσσών. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο πάρα πολλές πρεσβείες και πολιτιστικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων σχεδόν των χωρών της Ένωσης που εντάσσονται σε πολιτιστικές δράσεις και δίκτυα. Και αυτό το οποίο απαιτείται είναι ένας καλύτερος συντονισμός σε μια πρώτη φάση. Στα πλαίσια των προγραμμάτων τα οποία υπάρχουν, το θέμα της γλώσσας είναι κάτι το οποίο θα επιλέγεται από τις αντιπροσωπείες είτε της Ένωσης είτε των κρατών μελών που συμμετέχουν στις διαφορετικές πρωτοβουλίες. Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Βερζά σχετικά με τις μειονότητες. Πράγματι οι μειονότητες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να αγνοηθούν είναι χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο σεβασμός των μειονοτήτων. Τώρα για τον τίτλο έχω ήδη μιλήσει. Σίγουρα υπάρχει το θέμα και των πολιτιστικών ακολούθων και το πώς θα λειτουργήσουν στο μέλλον στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Τώρα το τι ακριβώς θέλουμε που είπε η κυρία Χόνιμπαλ Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι βασικός μας στόχος είναι η προώθηση της ποικιλία της Ευρωπαϊκής. Είναι ένα μέσο που συντονίζει τα υπάρχοντα μέσα, δεν δημιουργείται ένα νέο μέσο θα έλεγα, απλά προσπαθούμε όλα αυτά να λειτουργούν συνεκτικά και στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας να συνειδητοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συντονίζονται μεταξύ τους τα μέσα αυτά. όχι να λειτουργήσουμε σαν την αμερικανική μουσική βιομηχανία όπως είπαν ορισμένοι, αλλά να προωθήσουμε γενικά τα πολιτιστικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κύριος Μικαέλς και αναφέρθηκε και αυτό στα θέματα του τίτλου. Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση ειδικά μετά την, το κλείσιμο της συνεδρίασης για το τι ανησυχίες υπάρχουν για τον τίτλο. Συμφωνώ ότι οι λέξεις πολλές φορές έχουν στρατηγική σημασία. Η κυρία Πάκα, όπως είπα στην αρχή, είπε αυτά τα οποία ήθελα και εγώ να πω. Addressed a few of the issues regarding the concern for the lack of diversity, but και έτσι καλύπτονται και τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν σχετικά με τις φόβους για το μη σεβασμό της ποικιλία και της διαφορετικότητας. Μία μικρή ερώτηση. Πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Θα σας τα πω εγώ, μην ανησυχείτε, λέει η Πρόεδρος. you have it? Ah, before Πρώτα όμως, ο εκπρόσωπο, δείχνει όμως έναν ευρωβουλευτή, ο εκπρόσωπο τη Επιτροπής. Πού είναι ο κ. Κανία. Α, είναι από αυτή τη μεριά. Ναι, ναι, α, μάλιστα, εντάξει. Είναι από την άλλη. Μα ε, εκεί κανονικά κάθεστε. Α, θέλετε να κάθεστε δίπλα στη συνάδελφό μα μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Κατά σύμπτωση περισσότερο έχω καθίσει εδώ. Κανονικά θα έπρεπε κάθομαι απέναντι, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάντως που μας προσκαλέσατε. Ευχαριστώ επίσης για την μακρά και ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής σας. Σημείωσα προσεκτικά τα σχόλιά σας. Σε αυτή την πρώτη φάση, εγώ θα ήθελα να συνεργαστώ με την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ. Ε, εύχομαι να καρποφορήσει η συνεργασία σας αυτή. Τώρα, μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει στις 26 Δεκάτου. Υπάρχει σχέδιο, ρωτάει η Πρόεδρος. Όχι. Στις 26 Οκτωβρίου θα ξανασυζητήσουμε την κυρία Σχάκε. Ακόμη δεν θα υπάρχει όμως κείμενο. Ίσως όμως μπορεί να μας δώσει ένα πρώτο δομημένο σχέδιο. Στις 18 Νοεμβρίου θα υποβάλει το κείμενό της. 18 Νοεμβρίου. Η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιανουάριο πλέον στην Επιτροπή Πολιτισμού. Άρα θα υπάρχει χρόνο σίγουρα μέχρι αρχάς Δεκεμβρίου για κατάθεση τροπολογιών. Από τις 18 Νοεμβρίου και μετά, δεν ξέρω ακριβώς μέχρι πότε, τον Δεκέμβριο, θα δούμε και πόσο χρειάζεται για τη μετάφραση. Πάντως κάποια στιγμή αρχάς Δεκεμβρίου θα είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, η ψηφοφορία όπως είπα τον Ιανουάριο δεν, δεν, είναι και, δεν είναι και κατεπηγόν το θέμα. Βλέπετε πόσο αργά προχωρεί αυτή η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, άρα εμείς μάλλον θα είμαστε πολύ ταχύτεροι από αυτούς. Ε, άλλωστε οι πρέζεις μέχρι να λάβουν τα καθήκοντά τους, ου, θα αργήσουν ακόμη. Πιο πολύ είναι για... Τέλος πάντων δεν κάνω τα σχόλια αυτά, για ως πρόεδρος δεν επιτρέπεται. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ αγαπητοί Σχάκε, ήταν εξαιρετική συζήτηση πράγματι. Νομίζω ότι με την συνεργασία όλων η συζήτηση και η έκθεση θα είναι εξαιρετικές. Τώρα, ερχόμαστε σε ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα. βελτίωση δηλαδή, τη συμμετοχής των σπουδαστών στο πρόγραμμα Έρασμος. Μία ερώτηση. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί την ε, έχασα. Μα, μα το είπα, αρχές Δεκεμβρίου. 20, 20. 23 Οκτωβρίου, απαντά η κυρία Πακ, χωρίς να, ξέρουμε, χωρίς να έχουμε ακούσει την ερώτηση. Όχι, Σεπτέμβριο. Πες μου, έλα. Μια στιγμή σας παρακαλώ. Όπως είπα, 23 Σεπτεμβρίου. 23. Το μεσημέρι. Στις 12, ε. Καλά λοιπόν. Θα έρθουμε τώρα στην παρουσίαση του Ολλανδικού Πανεπιστημίου του ΕΝΤ. Εσείς παρακαλώ, ο κύριος της Κομισιόν και η κυρία των Φιλελευθέρων. Προσέξτε παρακαλώ τι λέμε. Είχαμε αναθέσει μία έρευνα για να δούμε ποια είναι, ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που είτε εμποδίζουν είτε οθούν τους ε, σπουδαστές να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Έρασμος που γνωρίζετε ότι λειτουργεί ήδη από το 1987 και είναι από τα πιο σημαντικά μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό και αυτό μας ενδιαφέρει να μάθουμε γιατί δεν ενδιαφέρονται περισσότεροι να συμμετάσχουν. Αν υπάρχουν παράγοντες που τους εμποδίζουν, αν είναι δυνατόν να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, απευθύνω θερμό χαιρετισμό στον καθηγητή Βόσενστάιν, που είναι συντονιστής έρευνας στο Πανεπιστήμιο αυτό των κάτω, των κάτω χωρών και θα παρουσιάσει σύντομα την έρευνα, η οποία εν συνόμψη περιλαμβάνεται στους φακέλους σας και βέβαια μετά την παρουσίασή του θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Παρακαλώ κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου και λοιποί παρόντες, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ για να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης μελέτης για τη λειτουργία του προγράμματος Εράσμους συμμετείχα σε μια πολύ ζωηρή συζήτηση και προηγουμένως και είδα πώς λειτουργεί η Επιτροπή σας στην πράξη. Να ευχαριστήσω και το Τμήμα Πολιτικής B, γιατί είναι αυτό το οποίο ζήτησε την εκπόνηση αυτής της μελέτης. Θεωρώ ότι το Εράσμις είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την διάδοση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών αλλά και οικονομικών διαστάσεων στην Ευρώπη. Έχουμε ένα-δύο τεχνικά θεματάκια να ρυθμίσουμε πριν μπορέσετε να δείτε τη μελέτη στις οθόνες σας. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από μια κοινοπραξία ερευνητικών ομάδων, σε μία από τις οποίες συμμετέχω κι εγώ, στις κάτω χώρες, αλλά ε, συνεργαστήκαμε και με διεθνείς εταίρους, όπως για παράδειγμα το Κέντρο ε, για την Ανώτατη Εκπαίδευση στο ΜΠΑΘ, ε, το ICEM και με το Anderson Elfers Felix. Τα λύσαμε τα τεχνικά θέματα, οπότε έχετε τις διαφάνειες. Στόχος λοιπόν της μελέτης ε, ήταν αυτά τα οποία εξήγησε ήδη η Πρόεδρος νομίζω. Θα σας πω κι εγώ ένα-δυο πράγματα τα οποία ε, έχουμε στη μελέτη μας. Έχετε ένα αντίγραφο της μελέτης όλης και η ε, σύνοψη θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες εξ όσων ενημερώθηκα. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον υπάρχουν οικονομικοί ή άλλοι φραγμοί που παρεμποδίζουν την συμμετοχή στο πρόγραμμα Εράσμου. Ποιοι είναι δηλαδή οι παράγοντε που μπορεί να περιορίσουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Εράσμου, διότι υπάρχουν κάποιε φήμε ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών στη συμμετοχή τους και στι ε, σπουδέ τους στο εξωτερικό ε, μπορεί να μειώνεται. Ισχύει βέβαια για κάποιες χώρες αυτό, δεν ισχύει για όλες τις χώρες. προσπαθήσαμε να απαντήσουμε ερωτήσεις για το τρέχον επίπεδο κινητικότητα στην Ευρώπη, κατά πόσον υπάρχουν οικονομικοί φραγμοί για τη συμμετοχή στο Εράσμου, είναι προσβάσιμο το Εράσμου ε, σε φοιτητέ από όλες τις κοινωνικο οικονομικέ ομάδες, ε, άτομα από κατώτατα επίπεδα μόρφωσης ή οικονομική κατάσταση σε σχέση με άλλους Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συμμετοχή, παραδείγματο χάρη το κατά πόσον ε, γνωρίζει κάποιος το πρόγραμμα Εράσμου, το κίνητρα των φοιτητών και φυσικά τι μηχανισμοί μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή στο Εράσμου. Πώς μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε τον αριθμό των φοιτητών που συμμετέχουν στο Εράσμους, διότι έχουμε ε, πολύ μεγάλους ε, φραγμούς, όχι μόνο για το Εράσμους, αλλά για την κοινωνικότητα εν γέννη στην Ευρώπη. Προκειμένου να εκπονήσουμε τη μελέτη λοιπόν, Ακολουθήσαμε την ε, εξή μεθοδολογία. Καταρχάς εξετάσαμε τι βιβλιογραφία υπάρχει για τη λειτουργία του Εράσμους, τι στοιχεία μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς από αυτό και ποια είναι τα εφιστάμενα στατιστικά στοιχεία. Προσπαθήσαμε επίσης να διευκρινίσουμε λίγο περαιτέρα τα ερωτήματα που θέλαμε να θέσουμε ε, μέσω μιας έρευνας. Μία έρευνα η οποία έγινε σε περιορισμένο αριθμό χωρών λόγω των χρονικών περιορισμών που είχαμε για την ε, περάτωση της μελάτης. Το 2006 είχε γίνει μια μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα. Εμείς λοιπόν ε, κάναμε κάποιες επιπρόσθετες ερωτήσεις ε, στα όσα ήδη γνωρίζουμε. Κάναμε λοιπόν μια μελέτη σε 7 χώρες, στην Τσεχία, στη Φιλανδία, στη Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχικώ είχαμε πρόθεση να συμπεριλάβουμε και τι κάτω χώρε, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να απευθυνθούμε σε φοιτητέ εκεί, διότι έχουμε πολύ μικρό αριθμό φοιτητών σε διάφορες κατηγορίες και τελικώς τους αποκλείσαμε από την τελική μας ανάλυση. Συνολικώς ε, είχαμε ε, πάνω από 21.000 απαντήσεις, σημαντικός αριθμός, συμπεριλαμβανομένων και φοιτητέ που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εράσμου, περίπου το 1 τρίτο εξ αυτών δεν συμμετείχαν. Θα εξηγήσω αργότερα και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που έχουμε που διαφοροποιεί τη μελέτη αυτή από άλλε μελέτε που έγιναν για το Εράσμου. Είχαμε κάποιου φοιτητέ οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο Εράσμου που απάντησαν στο ερευνητολόγιο και κάναμε και κάποιε πιο λεπτημερέ μελέτε σε τέσσερι χώρε: στη Φιλανδία, στι κάτω χώρε στην Πολωνία και στην Ισπανία. Εκεί μιλήσαμε σε εκπροσώπου Υπουργεία, σε μορφωτικών ιδρυμάτων ε, και έγιναν και κάποιες ε, ομάδες ε, μελέτης. Όπως σας είπα λοιπόν, το προστιθόμενο όφελος αυτής της μελέτης είναι να επικυρώσουμε τα αποτελέσματα που είχαμε βρει σε προηγούμενες μελέτες, να δούμε κατά πόσον υφίστανται ακόμα τα ίδια στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, ε, να κάνουμε μία νέα μελέτη φοιτητών, η οποία θα περιλαμβάνει και φοιτητές που δεν συμμετείχαν στο Εράσμους, αυτό είναι το νέο στοιχείο, τα κίνητρά του και τον τρόπο που το αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους οι μη στο και γιατί δεν συμμετείχαν ή γιατί να συμμετάσχει κάποιος. Και φυσικά είχαμε και τις πιο εις βάθος μελέτες, οι οποίες μας δίνουν κάποιες ε, πτυχές ε, ε, και από πλευράς ενδιαφερομένων. Τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία που διαπιστώσαμε. Καταρχάς ως προς την κινητικότητα. Δεύτερον, ω προ του ε, οικονομικούς περιορισμούς, ε, την εμπειρία των φοιτητών, ε, τα στοιχεία που μας υπέδειξαν οι φοιτητέ και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι και κάποια άλλα στοιχεία. Και τέλο θα καταλήξω σε κάποιες συστάσεις για το εράσμο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει μια συνεχής αύξηση στη συμμετοχή στα προγράμματα Εράσμου. Ωστόσο, το ποσοστό των φοιτικών που είναι ενεργοί στο εράσμος είναι περίπου 4% αν συνυπολογίσουμε και τους φοιτητές που έρχονται σε επαφή με το πρόγραμμα εράσμου σε όλη την ε, πανεπιστημιακή τους πορεία, στην εκπαιδευτική τους πορεία έχουμε ένα ποσοστό μεταξύ 1 και 1,5% αν λάβουμε υπόψη και φοιτητέ που συμμετέχουν στο σύστημα 4-5 χρόνια, τότε φτάνουμε στο σύνολο του 4% που σας ανέφερα. Η συμμετοχή είναι χαμηλότερη στα νέα κράτη-μέλη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 και μετά, αλλά εκεί αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα η συμμετοχή στο εράσμος. Οι λόγοι για την κινητικότητα είναι κυρίως ε, προσωπική εξέλιξη, ε, να αναπτύξει κάποιος τις προσωπικές του δεξιότητες. Ε, τώρα, τα ωφέλη από οικονομικής πλευράς και από πλευράς καριέρας δεν είναι ο βασικός στόχος ενός φοιτητή που συμμετέχει στο Εράσμος. Ναι, μεν αναφέρεται, αλλά δεν θεωρείται η προτεραιότητα και οι φοιτητέ Εράσμου κυρίως προέρχονται από ε, υψηλότερες ε, ομάδες από οικονομικής πλευράς. Ε, αυτό δεν θα εκπλήξει κανέναν, γιατί αν δούμε τη γενικότερη συμμετοχή στην ανώτερη, ανώτατη εκπαίδευση, αυτή είναι η τάση. Αν δούμε από εκεί και πέρα τα διεθνή στοιχεία, περιορίζεται ακόμα περισσότερο λόγω οικονομικών παραγόντων η συμμετοχή στο Εράσμου. Τουλάχιστον σε κάποιε χώρε, όχι παντού. Επίσης υπάρχει μια τάση οι φοιτητές να έρχονται από τα ε, παραδοσιακά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Υπάρχει μια εξαίρεση στη Φιλανδία όπου έχουμε και συμμετοχή από άλλους τομείς, κυρίως από φυσικές επιστήμες, αλλά η τάση είναι να, ε, είμαστε, να ε, προέρχονται από τα παραδοσιακά ακαδημαϊκά ιδρύματα και κυρίως από τις μεγαλύτερες πόλεις. Εδώ έχετε ένα χάρτη που δείχνει ε, τη αποσοστά εσωτερικής κινητικότητας, ε, ποιες χώρες ε, εισάγουν ή εξάγουν φοιτητές Εράσμους. Ε, το μπλε, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή και η Σουηδία, οι κάτω χώρες, η Δανία, είναι χώρες εισαγωγής φοιτητών Εράσμους. Οι βαλτικές χώρες που είναι πιο πολύ στο ροζ, είναι χώρες εξαγωγής ε, φοιτητών Εράσμους, που σημαίνει ότι υπάρχει μία ανισορροπία. Και αν θέλουμε να αυξήσουμε την κινητικότητα Εράσμους, οι χώρες οι οποίε εισάγουν ε, φοιτητέ θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρον στόχο, γιατί φαίνεται να προσελκύουν πολύ περισσότερους ε, φοιτητέ από όσου στέλνουν στο εξωτερικό. Και ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον ε, από πλευράς φοιτητών εκεί να μεταβούν στο εξωτερικό. Επίσης, μα ζητήθηκε να εξετάσουμε την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των φοιτητών. Μπορούμε να κάνουμε κάτι από αυτού. Η πρώτη ένδειξη που έχουμε είναι ε, μία αντιπαράθεση που κάναμε μεταξύ πλουσιότερων και λιγότερο πλούσιων χωρών. Αν το κατακεφαλή είναι ΑΕΠ, δηλαδή έχει σχέση με το ΑΕΠ, ε, με το Εράσμους και αν οι, φοιτητέ ε, οι φοιτητές από χώρες που είναι πλουσιότερες συμμετέχουν στο Εράσμους περισσότερο δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο σοβαρό συμπέρασμα. Τα ποσοστά των φοιτητών που συμμετέχουν στο Εράσμους ποικίλουν ε, ανάλογα με τη χώρα και αυτό βέβαια που θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε εδώ στο διάγραμμα είναι ότι οι χώρες που έχουν χαμηλότερο κατακεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση στους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εράσμους. Δηλαδή, στα νεότερα κράτη-μέλη, οι χώρες οι οποίες έχουν χαμηλότερο ΑΕΠ, μεταξύ 2004 και 2008, είχαν ένα ε, σημαντικό ποσοστό αύξησης ε, της συμμετοχής, ενώ στις ε, πλουσιότερες χώρες είτε είναι ε, σταθερό το ποσοστό είτε μειώνεται. Και εδώ έχετε το ενδιαφέρον ερώτημα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω καταλήλως, αλλά έχω μία σειρά από στοιχεία που θα μπορούσαν ίσως να μας οδηγήσουν σε κάποιο δίκτυ. Τα βασικά στοιχεία που διαπιστώσαμε ως προς τους, ε, ε, τα οικονομικά εμπόδια για τη συμμετοχή στο Εράσμος. το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι τα οικονομικά προσκόμματα είναι το βασικό εμπόδιο για τη συμμετοχή των φοιτητών στο Το 57% των φοιτητών που δεν συμμετέχουν στο Εράσμους θεωρούν ότι οι σπουδές στο εξωτερικό είναι πολύ ακριβές. Και το 29% απορρίπτει ε, το πρόγραμμα Εράσμους γιατί θεωρεί ότι η υποτροφία που λαμβάνει είναι πάρα πολύ μικρή και δεν μπορεί να καλύψει το κόστος της διαβίωσης στο εξωτερικό. Το κόστος και το επίπεδο της υποτροφίας ε, δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει τόσο. Θέλουμε να δούμε ε, τι ισορροπία υπάρχει μεταξύ των, ε, της σχέσης κόστους-οφελίας. Δηλαδή, εκεί μπορεί να υπάρξει το εμπόδιο. Θέλουμε να έχουμε μια ισορροπία, διότι υπάρχει πάντα το ερώτημα τι θα αποκομίσω εγώ αν μεταβώ στο εξωτερικό για να σπουδάσω, θα έχω καλύτερη καριέρα, θέσεις εργασίας κλπ. Σε χώρες που έχουμε υψηλή κινητικότητα, το ε, φαινόμενο της αγοράς εργασίας φαίνεται να μειώνεται. Ε, φοιτητές ε, που ε, συμμετείχαν στο Εράσμου στο παρελθόν είχαν υψηλότερους μισθούς ή πιο ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας, αλλά φαίνεται να υπάρχει μία μείωση αυτή τη στιγμή βάσει βιβλιογραφίας. Και η επίπτωση λοιπόν εδώ είναι ότι η προστεθέμενη αξία του Εράσμου για τους φοιτητές των συγκεκριμένων χωρών δεν είναι πλέον τόσο σημαντική και συνεπώς δεν θεωρούν ότι το εράσμος είναι επένδυση πλέον, είναι μια πολυτέλεια, κάτι επιπλέον και εφόσον είναι κάτι επιπλέον, οι φοιτητέ από τις χαμηλότερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες μάλλον δεν θα συμμετάσχουν, διότι θεωρούν ότι η επιπλέον προσπάθεια που πρέπει να γίνει, προκειμένου να πάει κάποιο στο εξωτερικό να σπουδάσει, το επιπλέον κόστος που υπάρχει, οι δυνητικές καθυστερήσεις ε, στο πτυχίο του στη συνέχεια. Όλα αυτά έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και είναι πιο σημαντικά από το οικονομικό θέμα. Κάποια άλλα στοιχεία που διαπιστώσαμε που σχετίζονται με τους οικονομικούς φραγμούς είναι η προθυμία να συμμετάσχει κάποιος ε, στο Εράσμους ε, που ε, σχετίζεται και με το ποσό της υποτροφίας αλλά και με τις αβεβαιότητες ως προς το κόστος να, σπουδάσει κάποιος στο εξωτερικό. Πόσο κοστίζει να νοικιάσω ένα δωμάτιο και πρέπει να κρατήσω και το φοιτητικό μου δωμάτιο στην άλλη χώρα, οπότε θα διπλασιαστεί το κόστος. Ε, μετά, το επίπεδο τη υποτροφία. Πόσα χρήματα θα πάρει υποτροφία. Υπάρχει διαφορά ανά χώρα, υπάρχει διαφορά ανά πανεπιστήμιο. Ε, πώς είναι το πρόγραμμα των πληρωμών. Πότε θα τα λάβω αυτά τα χρήματα. Στη συνέχεια στη μελέτη είδαμε κατά πόσον μπορεί να υπάρχουν και άλλοι φοιτητέ που ενδιαφέρονται με να ε, σπουδάσουν στο εξωτερικό, αλλά προς το παρόν δεν έχουν συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα Εράσμου. Και εξετάζοντα τα στατιστικά στοιχεία αυτών που δεν συμμετέχουν και που δεν ενδιαφέρονται γιατί είναι πολύ ψηλό το κόστος ή έχουν απορρίψει την ε, υποτροφή εράσμου, ε, υπολογίζουμε ότι έχουμε ετησίως περίπου 980.000 ε, με 1,5 εκατομμύριο φοιτητές που μπορεί να, ήταν, να, ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στο Εράσμος. Είναι τεράστιο λοιπόν το ποσοστό αυτό και δεν ε, μπορούμε να τους ε, αντιμετωπίσουμε. Δεν λέω ότι σίγουρα θα συμμετέχουν στο Εράσμος, αλλά υπάρχουν δυνατότητες. Επίσης, εξετάσαμε τα εθνικά συστήματα φοιτητών, κυρίως για τους φοιτητές που σπουδάζουν στη χώρα τους και κατά πόσον οι δυνατότητες που έχουν ε, να μεταβούν στο εξωτερικό ε, μπορεί να προκύψουν από κάποια επιπλέον κονδύλια, εάν δηλαδή φοιτητέ που μπορεί να σπουδάζουν με δικά τους έξοδα και όχι με έξοδα των γονιών τους, ε, μπορεί να επηρεάσουν τη συμμετοχή τους στο Εράσμους, δηλαδή το να είναι κάποιος οικονομικά ανεξάρτητος. Επίσης υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν επιπλέον υποτροφίες ε, για φοιτητέ που θέλουν να μεταβούν στο εξωτερικό. Ε, δεν καλύπτεται επιπλέον κόστος, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει το πόσο σημαντικό είναι να μετακινείται κάποιος. Δηλαδή, να λέμε ότι για το πανεπιστήμιό σας είναι σημαντικό το να μεταβεί κάποιος στο εξωτερικό και εκεί δημιουργείται διαφορετική νοοτροπία και στους φοιτητές. Επίσης, εξετάσαμε άλλα δυνητικά εμπόδια για τη συμμετοχή των φοιτητών στο Εράσμους και τα εντάξαμε σε τέσσερις βασικές κατηγορίες καταρχάς οι προϋποθέσεις του προγράμματος Εράσμους, το κατά πόσο είναι συμβατή ανώτατη παιδεία και τα συστήματα στις δύο χώρες, ε, τα εξάμηνα, τα τρίμηνα, το τρόπος που λειτουργούν, ο προγραμματισμός. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία για το τι γνωρίζει κανείς για ένα πρόγραμμα Εράσμους. Εδώ βέβαια έρχονται και οι προσωπικοί παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο. Κάποιοι δεν θέλουν να φεύγουν από την οικογένειά τους, κάποιοι επιθυμούν ακριβώς το αντίθετο κτλ. Υπάρχουν πολλά ε, προσωπικά διαφοροποιητικά στοιχεία. Από τις μελέτες που κάναμε μέχρι τώρα, το 24% των φοιτητών δεν ενδιαφέρονται σε καμία περίπτωση να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Είμαι στη χώρα μου, μια χαρά είμαι, δεν πάω πουθενά. Το 25%, 24%. το 34% δεν κινούνται, δεν είναι κινητικοί, γιατί φοβούνται ότι ε, τα πιστοτικά σημεία τους, δηλαδή τα credits, εν πάση περιπτώσει τα πανεπιστημιακά, δεν θα γίνουν αντικείμενο αναγνώρισης. Αυτό παραμένει εμπόδιο σε πάρα πολλές χώρες. Πάρα πολλοί φοιτητέ αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αμοιβαία αναγνώριση των μαθημάτων τα οποία θα κάνουν στις διάφορες σχολές. Το 62% των φοιτητών θέλουν να επιλέξουν ένα, όργα, ένα ίδρυμα πανεπιστημιακό εκτός του καταλόγου που καλύπτεται από το Εράσμος. Δεν είναι λοιπόν πάντα εύκολο για αυτούς. Το 41% των φοιτητών φοβούνται ότι έχουν ιδιαίτερα χαμηλές γλωσσικές ικανότητες για να αντιμετωπίσουν με το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών σε μια ξένη χώρα. ένα ποσοστό 46% δεν μετακινούνται για προσωπικούς λόγους και οικογενειακούς λόγους, 53% θέλουν καλύτερες ε, πληροφορίες για το Εράσμος και 35% πιστεύουν ότι έτσι όπως είναι σήμερα το Εράσμος δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο διοικητικό βάρος και σε επίπεδο πανεπιστημίου, εθνικό επίπεδο, διεθνές επίπεδο, εν πάση περιπτώσει πιστεύουν ότι η τεράστια διοικητική προσπάθεια και δεν θα την αναλάβουν. Υπάρχει επίσης μια σημαντική ομάδα των φοιτητών που πιστεύουν ότι το Εράσμους είναι κάτι το κοινωνικό και όχι τόσο πανεπιστημιακό. Πηγαίνει κανείς να σπουδάσει στο εξωτερικό γιατί είναι ωραία, είναι αστεία, γνωρίζει κόσμο και κάνει καλά πράγματα. και αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα σε σχέση με τον σοβαρό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις πανεπιστημιακές τους σπουδέ. Το 33% των φοιτητών έχουν κάποιες αβεβαιότητες σχετικά με το σύστημα εκπαίδευσης το οποίο πάνε να ενταχθούν. Δεν ξέρουν πού ακριβώς θα πάνε, πώς θα εγγραφούν, πρέπει να πληρώσουν, δεν πρέπει θα είναι στα αγγλικά, στα γαλλικά, σε άλλη γλώσσα. Υπάρχει επίσης και μία έλλειψη συνεκτικότητας ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα. Δεν εντυπωσιάζει κανέναν αυτό, γιατί αν δει κανεί τους φοιτητές οι οποίοι σε ένα εθνικό επίπεδο αποφασίσουν να ξεκινήσουν κάποιες σπουδές, Ξέρετε ότι το 30% μετά από το πρώτο έτος αναγκαστικά πηγαίνει σε κάτι άλλο, αλλά αυτό ισχύει για κάποιες χώρες. Και υπάρχει επίσης και σοβαρή ανησυχία για την ποιότητα του συστήματος της εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Κάποιοι παράγοντες οι οποίοι δεν θεωρούνται πολύ σημαντικοί είναι ε, η διάρκεια της επίσκεψης και του προγράμματος το οποίο θα παρακολουθήσουν Κάποιοι από τους φοιτητές έχουν ένα, μια δουλειά part-time και δεν θέλουν να την αφήσουν, αλλά εν πάση δεν είναι σημαντικός παράγον, δεν είναι μείζον εμπόδιο που θα τους αποτρέψει από το να πάνε στο εξωτερικό. Η έλλειψη προγραμμάτων στα αγγλικά δεν είναι σημαντικό πρόβλημα, γιατί πολλοί ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τα μαθήματα σε άλλες γλώσσες και υπάρχει επίσης και η έλλειψη υποστήριξης στα πλαίσια των φοιτητικών υπηρεσιών. Το τελικό κομμάτι είναι οι συστάσεις αυτής της μελέτης. Φαίνεται ότι υπάρχει πάντα μια μεγάλη ανάγκη για ακόμα περισσότερες υποτροφίες εράσμους. Υπάρχει δηλαδή ένα αρκετά μεγάλο δυναμικό το οποίο δεν έχει καλυφθεί. Και φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για να καλύψουμε την ζήτηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με τη σημασία των εμποδίων ανάμεσα σε χώρες. Αυτές ε, οι διαφορετικές μορφές εμποδίων που υπάρχουν για τους φοιτητές μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα νούμερο κάνει για όλους δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και υπάρχει επίσης μεγαλύτερη ανάγκη για να υπάρχουν και ε, σπουδές έρασμος και σε εθνικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς, σαν παράδειγμα, σε μία χώρα, στο εσωτερικό ε, μίας χώρας και δεν υπάρχει και σωστή ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενημερώνουν για τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Υπάρχουν και χώρες με υψηλή συμμετοχή οι οποίες υποφέρουν αυτή τη στιγμή από στάσιμους προϋπολογισμούς. Υπάρχουν λοιπόν τρεις επιλογές. Είτε να μειώσουν την ε, υποτροφία που δίνουν στους φοιτητές ή να απογοητεύσουν ένα μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών ή να πάρουν επιπλέον εθνική χρηματοδότηση. Λίγες χώρες το κάνουν αυτό, γιατί πολλές από τις χώρες αυτές ε, έχουν προβλήματα σε επίπεδο εσωτερικό χρηματοδότησης των φοιτητικών σπουδών το να προσθέσουν στις δυσκολίες αυτές επιπλέον κόστος για τη διεθνοποίηση των σπουδών και την κινητικότητα είναι πολύ δύσκολο. Φαίνεται λοιπόν ότι σε ορισμένες χώρες ε, δεν δαπανάτε το σύνολο του προϋπολογισμού Εράσμους και θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε καλύτερο κεντρικό ε, συντονισμό θα έλεγα έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις για το πόσο θα ωφεληθούν οι φοιτητές επαγγελματικά από τις σπουδέ τους αυτές. Εμείς λέμε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να υπολογίσει κανείς το κόστος και το κέρδος, το όφελος σε επίπεδο επαγγελματικό. Ξέρουμε επίσης ότι σε ορισμένες χώρες έχει αυξηθεί το κόστος των σπουδών, το κόστος εγγραφής σε κάποια πανεπιστήμια και οι φοιτητέ είναι λογικό να μην θέλουν να επενδύσουν ε, σε σπουδές στο εξωτερικό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι το πρόγραμμα Εράσμους είναι ιδιαίτερα επιτυχές στο να κινητοποιεί ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ε, παίρνουν υποτροφίες και πηγαίνουν σε επιχειρήσεις, μέσω επιχειρήσεων. Εδώ θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να καλύψουμε ακόμα καλύτερα τις ανάγκες της οικονομικής των φοιτητών. Θα πρέπει να μιλήσουμε και τα λεγόμενα soft skills και την προώθηση των μακροπρόθεσμων ωφελημάτων από τέτοιου είδους ε, soft skills όχι βέβαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί αυτό είναι πολύ περίπλοκο και θα καταστήσει την διαχείριση και το βάρος της διαχείρισης του Εράσμους ε, πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να προωθήσουμε την κινητικότητα και στις λιγότερο ε, αναπτυγμένες περιοχές, γιατί ξέρουμε ότι κυρίως ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών προέρχεται από τις αστικές περιοχές και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα από τα περιφερειακά ταμεία ίσως εδώ. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε και καλύτερη πληροφόρηση σε σχέση με το κόστος της κινητικότητας. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι πανάκριβη η κινητικότητα. Ναι, αλλά πόσο ακριβή είναι. Ένα πρόγραμμα το οποίο είχε γίνει εξ ονόματος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της διαβίου κατάρτισης λέγει ότι έχουμε στοιχεία πλέον τα οποία θα καταστήσουν τις εθνικές στατιστικές πιο κατανοητές και έτσι οι φοιτητέ που θέλουν να γίνουν ακόμα πιο κινητικοί να γνωρίζουν τις διαφορές στο κόστος ή πολλές φορές τις μη διαφορές στο κόστος. Πολλοί πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι ακριβό και λένε δεν θα πάνε, αλλά τελικά μπορεί να δούνε προσεκτικά αν κοιτάξουν ότι το κόστος δεν μπορεί να είναι και τόσο ψηλό μερικέ φορές. Υπάρχει επίσης και πρέπει να υπάρξει μάλλον μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με το ύψος της υποτροφίας. πώς θα είναι και τι κόστος θα καλύψει από την αποστολή του στο εξωτερικό. Θα πρέπει επίσης ένα μεγάλο τμήμα του Εράσμους να δίδεται εκ των προτέρων, έτσι ώστε να καλύψει άρξη ε, της διαδικασίας αυτής και όχι να τα δίνουν από την τσέπη τους και να περιμένουν στο τέλος μετά. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία για τους φοιτητές να πληρώνουν, να πληρώνουν συγγνώμη, το κόστος και για τις μεταφορές και το κόστος για το πανεπιστήμιο όταν χρειάζεται. και θα πρέπει επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα μεταφοράς των συστημάτων εθνικής στήριξης των φοιτητών. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση, ε, σαν παράδειγμα αν μάθω την παραμονή που πρόκειται να φύγω, μάθω τα χίλια ευρώ ε, ότι θα πάρω μαζί μου χίλια ευρώ για να πάω σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, αυτό δεν είναι και τόσο πολύ χρήσιμο, αλλά αν είμαι σωστά ενημερωμένο, τότε μπορώ να προσθέσω τα 1.007 ευρώ στην υποτροφία Εράσμους και τότε να καταστεί η πιθανότητα μετακίνησης εφικτή. Ένα σημαντικό θέμα επίσης είναι το θέμα της αναγνώρισης των μαθημάτων. Νομίζω ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, για τη συμβατότητα των μαθημάτων και των credits των πανεπιστημιακών. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με φοιτητέ που πηγαίνουν σε άλλα πανεπιστήμια και δεν αναγνωρίζονται τα credits τα οποία παίρνουν σε διαφορετικές φάσεις. Και προσπαθούν να καταλάβουν από πριν τι ε, μπορεί να τους βοηθήσει στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουν για το Εράσμος. Η υποτροφή Εράσμους θα πρέπει επίσης ε, να αντιμετωπιστεί και στα πλαίσια των λεγόμενων διπλών διπλωμάτων. Γιατί όλο και περισσότερα είναι αυτά τα διπλά διπλώματα ανάμεσα σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Δύο πανεπιστήμια μεταξύ τους πολλές φορές αντιπροσωπεύουν ε, μια δυνατότητα καλύτερης αναγνώρισης και κατανόησης του τρόπου λειτουργίας και αναγνώρισης επίσης των credits τα οποία δίνουν και επίσης υπάρχει δυνατότητα και για μικρότερης χρονικής διάρκειας προγράμματα όπως θερινά πανεπιστήμια κτλ. Είναι διαφορετική αυτή η εμπειρία. Υπάρχει η δυνατότητα τέτοιων πανεπιστημίων θερινών ε, όπου είναι πολύ σημαντικές οι συναντήσεις αυτές ακόμα και αν κρατάνε μόνο μία εβδομάδα, μία ή δύο εβδομάδες πολιτιστικά τουλάχιστον, πολιτισμικά μάλλον να το πω καλύτερα, ωφελούνται οι φοιτητέ από αυτή τη μορφή της κινητικότητας. Και ίσως να αντιμετωπιστεί και το θέμα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Εράσμους για μεγαλύτερες χρονικές διάρκειες. Έρχομαι στην τελευταία διαφάνεια. Συστάσεις για την σωστή τοποθέτηση των προγραμμάτων στο εσωτερικό του Εράσμους να προσπαθήσουμε επίσης να βελτιώσουμε και τις δυνατότητες κινητικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί αν μπορούν οι καθηγητές και οι μαθητές στη δευτεροβάθμια να αποκτήσουν ένα άρωμα διεθνούς συνεργασίας και εμπειρίας, τότε ε, θα γίνουν πολύ πιο κινητικοί στο μέλλον. Εγώ συμμετέχω σε μια ένωση διευθυντών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στη χώρα μου, στην πόλη μου μάλλον, και συνεργαζόμαστε με την Ιρλανδία, κάνουμε κάποιες μικρές ανταλλαγές και έτσι τα παιδιά παίρνουν ένα άρωμα λοιπόν των δυνατοτήτων που υπάρχουν για τις, κοινο... για τις μετακινήσεις τους βλέπουν ότι υπάρχουν και άλλες χώρες λοιπόν εκτός από τη δική μας χώρα και σε μικρή ε, ηλικία. Και στη, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτό είναι κάτι το πολύ χρήσιμο. Θα πρέπει η προώθηση του προγράμματος Εράσμους να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ίσως δημιουργώντας κεντρικά πόρταλς ε, στο διαδίκτυο και δίδοντας ε, ε, μαθήματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Εράσμους για όλους τους πρωτοετής φοιτητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μαθαίνουν ακριβώς οι φοιτητές από την αρχή. Γιατί υπάρχει ένα 20% σχεδόν του πληθυσμού των φοιτητών που τελειώνουν τις σπουδές τους και που δεν έχουν πάρει είδηση ότι υπάρχει το Εράσμος και προφανώς εκεί μπορεί να υπάρχουν θέματα προκατάληψης που δεν επιτρέπουν τη σωστή ενημέρωση, αλλά εν πάση περιπτώσει η δουλειά υπάρχει και πρέπει να γίνει γνωστή. Επίσης, αν δεν θέλουμε να έχουμε μια ιδιαίτερα συγκεντρωτική αντιμετώπιση, ας ακολουθήσουμε την αποκεντρωμένη, αλλά ε, με ε, πολλές εθνικές δυνατότητες χρήσης του Εράσμους μέσω των βέλτιστων πρακτικών, μέσω των παλαιών μαθητών και φοιτητών που χρησιμοποίησαν το Εράσμος, μέσω ε, θα έλεγα σεμιναρίων για τα υπέρ και τα κατά της μετακίνησης των φοιτητών. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους φοιτητές, να μην κάνουμε τέτοια σεμινάρια θα έλεγα για τους φοιτητές που θα πάνε στο εξωτερικό αλλά για όλους τους φοιτητές έτσι ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τις δυνατότητες που έχουν και να αναγνωρίσουμε καλύτερα τα εθνικά δίκτυα Εράσμους. Ευχαριστώ λοιπόν, ελπίζω να φώτισα λίγο περισσότερο κάποια από τα θέματα σχετικά με το Εράσμος που να μην ήταν μέχρι τώρα ξεκάθαρα. Ελπίζω ότι το πρόγραμμα Εράσμος θα παραμείνει προτεραιότητα στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον. Αν έχετε ε, περισσότερες λεπτομέρειες. Για όλα αυτά έχετε ε, τα στοιχεία μου ε, και στο διαδίκτυο. Θα σας απαντήσω αμέσως στις ερωτήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική πραγματικά η παρουσίασή σας. And, Άνοιξε τα μάτια μας για ορισμένα πράγματα, αλλά επίσης επιβεβαιώνει και ορισμένες εμπειρίες μας. Μη λησμονείτε ότι έχουμε το πρόγραμμα Κομένιους, το οποίο δημιουργήθηκε το 1995, ειδικά επειδή θέλαμε να ενημερωθούν και τα παιδιά, όχι μόνο οι σπουδαστές, ότι η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος ενδιαφέρον περίπλοκος κόσμος και από την εποχή του τελευταίου προγράμματος εκπαίδευσης έχουμε τη δυνατότητα να πάνε στην Αλοδαπή για, για ένα χρόνο. Εντάξει, δεν ε, χρησιμοποιείται ακόμη πάρα πολύ, αλλά είναι μια αρχή. Θα πρέπει όμως πράγματι να ε, κινήσουμε το ενδιαφέρον του κοινού και στις χώρες μας. Και βεβαίως όχι μόνο οι σπουδαστές αλλά και οι καθηγητές. Αυτό λοιπόν ας είναι κάτι που θα ενδιαφέρει και τους καθηγητές. Και δεν είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζονται μετά τα πτυχία που αποκτούν μέσω του Εράσμου. Δεν ευθύνεται το πρόγραμμα για αυτό, ούτε εμείς, αλλά α, αυτός ο παραλογισμός αυτών των στενόμυαλων καθηγητών και εδώ και εκεί που δεν αναγνωρίζουν το τι γίνεται σε άλλες χώρες του κόσμου. Έτσι λοιπόν η διαδικασία της Μπολόνια, αν πρόκειται να έχει κάποια, αποτα... κάποια θετικά αποτελέσματα, αυτό θα πρέπει να είναι βεβαίως ένα από τα θετικά. Α, ο κύριος Μπερλινγκουέρ θα λάβει το λόγο, που βεβαίως και αυτός είναι μέσα στα πανεπιστήμια. Άλλωστε συναντηθήκαμε στην Πολόνια παλαιότερα, αν θυμάμαι καλά. Χαίρομαι που με μπερδέψετε με τον κύριο Βάτιμο. Κομπλιμέντο είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι ζήτησε αυτή τη μελέτη. Και φυσικά τα ερευνητικά ιδρύματα του ΤΣΕΠΣ επειδή έκανε αυτή την έρευνα, διότι είπε κάτι πολύ σημαντικό. Να σας διορθώσω, το Κοινοβούλιο τη ζήτησε αυτή τη μελέτη και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλο το Κοινοβούλιο, λέει ο κ. Μπερλιγκέρ. Α, συγγνώμη, εννοούσα την Επιτροπή. Δεν ήθελα να πάρει τα εύσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε. Συγγνώμη, η γλώσσα μου είναι φτωχή, λέει Επιτροπή και για τα δύο, ενώ εγώ εννοούσα την Επιτροπή μας και όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος πάντων, η μελέτη αυτή είναι σημαντική διότι αποκαλύπτει πόσο δύσκολο είναι σήμερα να έχουμε ευρωπαϊκή πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης το Εράσμους δεν είναι απλώς ε, μία μικρή στιγμή της ακαδημιακής καριέρας κάποιου. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι ευνοεί τον εξευρωπαϊσμό των πανεπιστημιακών σπουδών και επομένως και της αγοράς εργασίας ε, στα υψηλά επαγγέλματα ναι μεν υπάρχει αύξηση, αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες ε, στις οποίες ε, αρχίζει να παρουσιάζεται μείωση. Και υπάρχουν κάποιες χώρες ε, στις οποίες δεν καλύπτονται όλες οι θέσεις οι οποίες είναι στη διάθεση των φοιτητών. Επομένως, ελοχεύει ο κίνδυνος κρίσης. Τους λόγους τους ακούσαμε. Οι λόγοι είναι οι ίδιοι για τους οποίους ε, δυσχεραίνεται η διαδικασία της, της Μπολόνια. Ο ακαδημαϊκός κόσμος και οι χώρες μέλη δεν δέχονται πλήρως ε, την ε, διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των πανεπιστημίων. Επομένως το Εράσμους ουσιαστικά είναι ένα τυχαίο περιστατικό στην ακαδημαϊκή καριέρα ενός φοιτητή, ενώ θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών του. τι βοήθεια δίνεται πέραν της οικονομικής συνδρομής. Παραδείγματος χάρη, οι χώρες οι οποίες υποδέχονται φοιτητές, ε, τους ε, συνδράμουν ως προς τη στέγαση, το να τακτοποιηθούν, να ε, ενταχθούν στο πανεπιστημιακό βίο πλήρως ή τους αφήνουμε στη μοίρα τους. Το γεγονός ότι οι καθηγητές που στέλνουν τα παιδιά στο εξωτερικό και μετά δεν αναγνωρίζουν τις σπουδέ τους, διότι υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις τα ε, παιδιά μεταβαίνουν στο εξωτερικό και δεν αναγνωρίζονται. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή έλλειψη ευαισθησίας, διότι δεν αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι τμήμα του προγράμματος σπουδών του φοιτητή. Και αυτό είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει το απαραίτητο πρόγραμμα σπουδών, ώστε να υπάρχει μια προσέγγιση των προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ο καθένας κάνει τα δικά του, προχωράει μόνος του και η διαδικασία της Μπολόνια ε, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και φυσικά υπάρχει και μία εχθρική ε, εξ, εκστρατεία στον τύπο που είναι η ίδια εκστρατεία στον τύπο που παρουσιάζει το Εράσμος ως ένα άλμα στο κενό και φυσικά ε, την προωθεί αυτή τη συγκεκριμένη νοοτροπία. Στις Ιταλικές εφημερίδες κάθε μέρα διαβάζουμε η διαδικασία τη Μπολόνια απέτυχε. Καταλαβαίνετε με τι ε, ε, ψυχικά αποθέματα στέλνουν οι γονείς από εκεί και πέρα τους φοιτητέ να σπουδάσουν. Ότι υπάρχει αυτό το δράμα και φαίνεται ότι τα πανεπιστήμια και οι χώρες μέλη έχουν αφήσει τη διαδικασία αυτή στη μοίρα της και δεν την βοηθούν. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να ζητήσουμε είναι τόσο τα κρατημέλη όσο και ε, οι επικεφαλείς των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων να δεχτούν το Εράσμους ως κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείτε, το οποίο θα ε, το προβλέπουμε σε όλες του τις πτυχές και θα είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε τον αριθμό των φοιτητών. Το 4% των φοιτητών είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι χρειάζονται κονδύλια, αλλά δεν είναι τα πάντα θέμα χρημάτων όπω ακούσαμε στη μελέτη. Είναι διαφωτιστικό αυτό το έγγραφο, διότι μα λέει ότι κρυβόμαστε πίσω από το γεγονό ότι υπάρχει οικονομική κρίση και δεν υπάρχουν χρήματα, ενώ θα μπορούσαμε να λάβουμε μία σειρά από άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν από αυτή τη πλευρά και ε, το επαναλαμβάνω συνεχώ, αλλά είναι εξαιρετική έκθεση. Ε, για τον ίδιο λόγο δεν πολλαπλασιάζεται η αναγνώριση των ε, διπλών ε, πτυχίων, ε, διότι δεν υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, υπάρχει μια αντίσταση κατά του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και εμείς αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και η πρόταση που μας γίνεται εδώ μας βοηθά. Πρόκειται για ένα σημείο το οποίο ενδυναμώνει τις δράσεις μας. Ευχαριστώ κύριε Μπερλενγκέρ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ομιλητή και για μια ακόμη φορά συμφωνώ μαζί σας με τη γνώμη την οποία εκφράσατε για το ότι από τη μία μας ικανοποιεί το να βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση και σας ευχαριστώ όλους που δεχθήκατε την τροπολογία στον προϋπολογισμό γύρω από όλα αυτά τα θέματα, τα οικονομικά που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα αυτά και όχι μόνο το Εράσμους. Αντιδρώντας λίγο σε αυτά που είπε και ο κύριος Μπεβλινγκουέρ, να πω ότι θα πρέπει να μην αγνοήσουμε τις δυσκολίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν και τα εμπόδια τα οποία οφείλονται στις κυβερνήσεις των κρατών. Έχω εργαστεί στην έκθεση για τη διαδικασία της Μπολόνιας και για τη σχέση επιχείρησης πανεπιστημίου. Η διαπίστωση την οποία έκανα σχετικά με αυτά τα οποία συνέβησαν στη Γαλλία σαν παράδειγμα είναι ότι αν η γαλλική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει λιγότερο τη διαδικασία της Μπολόνια λέγοντας ότι είναι η αιτία για κάποια μέτρα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τη διαδικασία της Μπολόνια αλλά τα οποία έπρεπε να ληφθούν στη Γαλλία και τα οποία δεν άρεσαν στους φοιτητές και στους διδάσκοντες. Τα έριξαν όλα στην Πολόνια λοιπόν, ενώ ήταν αυστηρά εθνικά μέτρα, ε, απλά το έκαναν για πολιτικούς λόγους, οπότε πολιτική είναι και η ευθύνη. Ίσως επί τη βάση αυτής της μελέτης μπορούμε να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας, να βασιστούμε στις συστάσεις τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτά να τα αποφασίσουμε βέβαια στη συνάντηση των συντονιστών και για τον κύριο Βόζενστάιν. Διερωτώ με για τις ε, κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες και τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Γιατί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και εμπόδια, υπάρχουν όμως και πολιτιστικά εμπόδια. Ξέρετε ότι στις ε, ασθενέστερες οικονομικές κατηγορίες το να πάει κανείς στο εξωτερικό δεν έχει την ίδια σημασία και το ίδιο βάρος ε, με τις περιοχές οι οποίες έχουν ε, υψηλότερα εισοδήματα και αυτό γιατί οι περισσότεροι ε, μαθητές και φοιτητές από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα δεν πηγαίνουν ποτέ στο εξωτερικό. Ενώ όταν έχουν μεσαία προς υψηλά πηγαίνουν πολύ συχνά στο εξωτερικό. Θα πρέπει λοιπόν και ο πολιτιστικός παράγων να μην αγνοηθεί. Είπατε επίσης στην περίληψη που μας δώσατε στα γαλλικά, είδα ότι η Φιλανδία και η Σουηδία ήταν σε μια σχετικά διαφορετική θέση σε σχέση με την προώθηση αυτών των ανταλλαγών. Ξέρω ότι δεν ε, μπορείτε να μου δώσετε απάντηση τώρα γιατί έχουμε καθυστερήσει, αλλά να μου δώσετε μια γραπτή απάντηση. Αυτό σημαίνει ότι η φιλανδική και η σουηδική κυβέρνηση συνοδεύουν τα προγράμματα αυτά με τη δική του συμμετοχή. Αν δεν με καταλάβατε γιατί τα είπα βιαστικά θα σας τα στείλω και γραπτά. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έπρεπε να τελειώσουμε στις 12 παρατέταρτο. Έχουν άλλοι δύο ζητήσει το λόγο και γι' αυτό σας παρακαλέσω να είσαστε πάρα πολύ ε, σύντομοι. Μπόρις και Βάτιμο. να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη μελέτη σας, μια μελέτη η οποία σε βάθος κάνει θα έλεγα μια σωστή περιγραφή των εμποδίων αλλά και των εκτιμάτων του συστήματος αυτού. Και νομίζω ότι οι Υπουργοί Παιδείας θα, θα είχαν πολλά να κερδίσουν αν ε, διάβαζαν προσεκτικά αυτή την έκθεση realizowali na poziomie pobytu w ramach Erasmusa, a także na e, poziomie e, e, być może skojarzenia tego ze stypendiami. Συνεπώς, ο σύνδεσμος ανάμεσα στο πρόγραμμα Εράσμους και ε, τις εθνικές, τα εθνικά συστήματα υποτροφιών παρουσιάζει πολύ ε, ενδιαφέρον, όπως είπε λοιπόν και ο μιλητής, ο κύριος ομιλητής, αυτοί που ασχολούνται σε εθνικό επίπεδο στα διάφορα υπουργεία με τα θέματα αυτά θα κέρδιζαν πολλά διαβάζοντας την έκθεση. Να δούμε και ποιοι είναι οι ισολογισμοί ανάμεσα στους εξαγωγείς και εισαγωγείς σε εισαγωγικά φοιτητών, σε εισαγωγικά. Η Πολωνία είναι πιο εξαγωγική χώρα παρά εισαγωγική. Εγώ έχω μιλήσει με πολλούς φοιτητές οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα σε επίπεδο γλωσσικό, ακόμα και με την αγγλική γλώσσα. Εδώ είναι ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πω επίσης ότι παντού όπου τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν το σύνολο των πιστώσεων, τότε θα πρέπει να μεταφέρεται το υπόλοιπό τους στις χώρες οι οποίες είναι σε θέση να τις καταναλώσουν και να καλύψουν αυξημένη ζήτηση. Ένα άλλο θέμα το οποίο έθεσε ο κ. Φώσενστάιν είναι το νομικό θέμα. Γιατί τόσο λίγοι φοιτητέ ενδιαφέρονται στο κοινοτικό δίκαιο σαν παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο θέμα εικόνας. Eh, eh, Εγώ πάντα σκέφτομαι τι αρμοδιότητα έχουμε εμείς ως Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις επενδύσεις που κάνουν τα κράτη-μέλη για το Εράσμους, για τα πανεπιστήμια εν γέννη. Εξακολουθώ να μην το αντιλαμβάνομαι. Πριν από δέκα χρόνια ήμουν μέλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά, τότε γνωριστήκαμε κυρία Πακ Έλεγα απλώς να αυξηθούν ε, τα επιδόματα για τους Ιταλούς φοιτητούς τε. και ε, σκέφτηκα ότι δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι θέμα των κυβερνήσεων και θα ήθελα να γνωρίζω σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ε, σε επίπεδο κυβερνήσεων. Εάν γίνει έκθεση ίδια πρωτοβουλία, θα ήθελα να εμβαθύνουμε στο θέμα του ελέγχου και της αρμοδιότητας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπησέρχεται στα εθνικά θέματα για τα θέματα παιδείας. Κύριε Παλιαδέλη. 2009 uh, uh, Είχα καταθέσει το Δεκέμβριο του 2009 μια ερώτηση σχετικά με τη μείωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Εράσμος και πήρα μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση από τον κύριο Σεύκοβιτς. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας, μπορώ να σας τη δώσω αναγνωρίζει τα περισσότερα από τα αποτελέσματα στα οποία αναφερθήκατε κύριε Βόσενστάιν και υπόσχεται ότι σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο για το 2009 μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας θα επιληθεί το πρόβλημα. Διαρωτώ με λοιπόν, αυτοί στους οποίους θέσατε τις ερωτήσεις, τους φοιτητές τους οποίους ρωτήσατε. Ήταν αυτοί οι οποίοι φυσικά πήραν μέρος στο εράσμος, έτσι δεν είναι, πήγανες και πήραν μέρος στο εράσμος, έτσι δεν είναι. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιη, αλλά θέσατε το ερώτημα σε αυτούς οι οποίοι πήραν μέρος στο Εράσμος, γιατί αντίθετα από το οικονομικό πρόβλημα, νομίζω ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, το κοινωνικό και πολιτισμικό αποτέλεσμα της συμμετοχής στο Εράσμους είναι εξαιρετικά ισχυρός παράγων. Θα ήθελα λοιπόν να είχατε συμπεριλάβει ε, ε, και τις ιδέες αυτών που πήραν μέρος στο ε, Εράσμος παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Το έχει κάνει λέει η κυρία Πακ. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα, χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω η Επιτροπή σα για την κινητικότητα των σπουδαστών στον Έρασμο και εμείς ενδιαφερόμαστε βεβαίως ε, να αυξηθεί και η ποσότητα και η ποιότητα της κινητικότητας και ε, χαιρόμαστε για τη μελέτη που έχει γίνει που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της παρούσας Επιτροπής. Και εμείς είδαμε το 2008 και 2009 σημαντική αύξηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Εράσμος, ακόμα στις αρχές του προγράμματος NLP, τα επόμενα δύο χρόνια δεν πιστεύω ότι θα δούμε ρεαλιστικά άλλη αύξηση. Θα σταθεροποιηθεί ή θα υπάρξει ελάχιστη αύξηση. Συμφωνώ με τα συμπεράσματά σας, τις μελέτης δηλαδή, και επιβεβαιώνει παλαιότερα πορίσματα. Δεν βλέπω να έχουμε διαφορετική γνώμη προκειμένου. Υπάρχει και ένα μεγάλο ε, δυναμικό που δεν έχει εξαντληθεί ακόμη. Ο έρασμος λειτουργεί πολύ καλύτερα όταν υπάρχει μια διεθνοποίηση του, των πολιτιστικών. Και σε ό,τι αφορά τις συστάσεις θα τις εξετάσουμε με λεπτομέρεια αλλά από τα πιο σημαντικά που λέχθηκαν είναι ότι για να αντιμετωπιστεί το κοινωνικονομικό υπόβαθρο, αυτό πρέπει να γίνει κυρίως στο εθνικό επίπεδο. Και ένα θέμα ακόμη, το οποίο έχουμε ήδη σημειώσει εμείς, ίσως η μελέτη να υποτιμά τα ευεργετήματα του προγράμματος Έρασμος, που είναι πολύ μεγάλα για τους συμμετέχοντες. Και με την ανάλυση της μελέτης Βαλέρα, που δείχνουν ότι τα ευεργετήματα μεγαλώνουν και με τον χρόνο, και το feedback που έχουμε από τους σπουδαστέ που συμμετέχουν αλλά και από τους εργοδότες είναι ότι εκτιμούν ιδιαίτερα την ε, μετακίνηση αυτή των σπουδαστών στο εξωτερικό. Θα εξετάσουμε λοιπόν όπως είπα τις συστάσεις με ε, περισσότερες λεπτομέρειες και βέβαια για θέματα αναγνώρισης και προώθησης ε, της κινητικότητας με προγράμματα τα οποία σε δύο εβδομάδες το πολύ θα ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα τελευταίο συμπέρασμα είναι ότι όλες οι άλλες προσπάθειες που κάνουμε σε άλλους ε, τομείς ε, για την αντιμετώπιση δηλαδή, των διαφόρων φραγμών, τα οικονομικά θέματα είναι, εξακολουθούν, το οικονομικό θέμα εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό. Και θα χρειαζόταν για να υπάρξει αύξηση των συμμετεχόντων σημαντική αύξηση του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Λίγος χρόνος μας μένει. Πολύ, πολύ σύντομη απάντηση λοιπόν. Θα παρακαλέσω δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη της την έρευνα και να μας δώσει γραπτός απάντηση. Είναι δυνατόν αυτό? Συμφωνώ μαζί σας, θα αναλύσουμε αυτό το χρήσιμο έγγραφο και θα σας δώσουμε γραπτός απάντηση. Εσείς κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ όλους και όλους για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τα πραγματικά εξαιρετικά σημαντικά σχόλιά σας. Πώς συνδέεται το κοινωνικονομικό καθεστώς των σπουδαστών με την κινητικότητα. Φαίνεται ότι οι ασθενέστεροι οικονομικά ε, σπουδαστές σε πλουσιότερες χώρες συμμετέχουν λιγότερο στον έρασμο. Αυτό φαίνεται. Σε φτωχότερες όμως χώρες, τέτοιου είδους σπουδαστέ είναι πλέον πιθανό να συμμετάσχουν. Είναι λοιπόν εκεί οι αναλογίες πιο ισορροπημένες μέσα στο συνολικό αριθμό των φοιτητών. Δεν παρεμποδίζεται απολύτω λοιπόν η κινητικότητα από το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο, διότι οι φτωχότεροι ε, φοιτητέ από τι οχότερε χώρες πρέπει να κάνουν μια διπλά, διπλή προσπάθεια για να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Για αυτούς η κινητικότητα αυτή αποτελεί επένδυση, ενώ στις ε, παραδοσιακά κινητικές χώρες φαίνεται να είναι περισσότερο ένα είδος πολυτέλειας που προσφέρουν στον εαυτό τους. Αυτή είναι η ιδέα που βγαίνει, ε, που προκύπτει από τη μελέτη. Και αυτό θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένους από τους ερωτώντες. Και για παράδειγμα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι στην Σουηδία η χορήγηση παραπάνω κονδυλίων στο εθνικό επίπεδο ε, βοήθησε. Είναι λοιπόν και εθνική ευθύνη και θα πρέπει να λεχθεί στους ενδιαφερόμενους τι πράγματα, τι, τι, μπορούν, τι ωφέλη μπορούν να έχουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα. Η σας ευχαριστώ που υπήρξατε και σύντομο, Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ και εσά και του συνεργάτε σα, κύριε Βόσενστάιν, ε, για τη χρήσιμη αυτή μελέτη. Θα δούμε αν θα τη χρησιμοποιήσουμε ως βάση για μια έκθεση πρωτοβουλίας. Οι συντονιστές θα κληθούν να το κρίνουν. Υπάρχουν άλλα διάφορα θέματα. Οκ, λοιπόν, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου η επόμενη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ και θα...